Καλή σας μέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Προτείνω να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και πάλι. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους συναδέλφους των δύο επιτροπών, Ήτρα και Τραν. Θα έχουμε μία κοινή συνεδρίαση. Έχετε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρώ ότι μπορεί να εγκριθεί το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε απευθείας συνδεδεμένοι και θα από το ίντερνετ. Θα ήθελα και πάλι να καλωσορίσω τα μέλη των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών που θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για αυτό τον τόσο σημαντικό φάκελο του μηχανισμού συνδέοντας την Ευρώπη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το καλό πνεύμα συνεργασίας που επικρατεί μεταξύ των δύο επιτροπών και θα ήθελα να δώσω το λόγο αμέσως στην, στην κυρία Ντέλη, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα πριν να αρχίσουμε να συγχαρώ για την εκλογή του τον κύριο Μπουσόη. Θα δείτε πόσο ενδιαφέρουσα είναι η δουλειά του Πρόεδρου, αλλά τι φόρτο εργασίας σημαίνει αυτό για τον Πρόεδρο. Θα τον συγχαίρω λοιπόν και χαιρετίζω και τον κύριο Βάγνερ από το Τυρόλο που είναι πρόεδρο μέλος της Επιτροπής Περιφερειών που θα παρακολουθήσει τις συζητήσεις που θα κάνουμε. Σας καλασορίζω και πάλι. Προσκάλεσε κυρία Τελέρ. Πού είστε, πού είστε, δεν σας βλέπω. Α, σας είδα τώρα. Καλωσορίσατε και σας. Σήμερα αγαπητοί συνάδελφοι, θα ασχοληθούμε με το μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη. Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης εξαιρετικά σημαντικό για τον εξυγχρονισμό και τα στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και της ε, ψηφιακής τεχνολογίας. Οι δύο επιτροπές μας κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας συμμετείχαν για να μπορέσουν να καθορίσουν στον τομέα κλειδί αυτό σε πρώτη ανάγνωση τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιλαμβάνει μία μερική συμφωνία που έγινε μετά από διαπραγματεύσεις πάρα πολύ εντατικές με το Συμβούλιο και την Επιτροπή αλλά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εργασία αυτή εάν δεν έχουμε και τα ακριβή στοιχεία και κονδύλια του προϋπολογισμού. Δεν είναι έτοιμο το διαπραγματευτεί το Συμβούλιο. Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το σύνολο του PDP και δεύτερον, στα πλαίσια του ίδιου του μηχανισμού, στα πλαίσια της συναπόφασης και πριν να υιοθετήσει την απόφαση πρώτη ανάγνωση στο Συμβούλιο, πρέπει να συνεχίσουμε και ελπίζω ότι θα ολοκληρώσουμε τη μελέτη του φακέλου αυτού έγκαιρα, ώστε ότι ε, επόμενος μηχανισμός να είναι έτοιμος το 2021. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές. Κύριε Μαρινέσκου, είστε εδώ. Κύριε ρικέ που είστε. Ορίστε και πάλι να σας ευχαριστήσω. Και κυρία Βιρκούνεν, που είστε εκεί. Σα ευχαριστώ και πάλι και θα ήθελα να ευχαριστήσω και του και συζητητή για την έκθεση αυτή. Πρόκειται για πολύ και εκτενείς διαπραγματεύσει που κάνετε και σήμερα ήρθε η ώρα τη ψηφοφορία. Αποφασίζουμε λοιπόν σήμερα ποιο είναι το επόμενο στάδιο το οποίο θέλουμε να έχουμε για την απόφαση αυτή. Σύμφωνα με του κανόνε που είναι πάρα πολύ σαφεί, προβλέπονται διαπραγματεύσει early second reading, σύμφωνα με το άρθρο 72 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα εργαστούμε για τις περίφημες διαπραγματεύσεις μας έχουν ατεθεί, δηλαδή πρώτα απ' όλα μη με κοιτάς έτσι, Κάρε. Μη με κοιτάς έτσι, λέει η Πρόεδρος. Έτσι όπως εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, η απόφαση διαπραγματεύσεις απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των δύο επιτροπών. Οι δύο επιτροπές από κοινού αποτελούνται από 120 μέρη, άρα η απόλυτη η πλειοψηφία είναι 61 μέλη. Για να οργανωθούμε σωστά για την ψηφοφορία, θα σας ζητήσω πρώτα απ' όλα να δείτε εάν έχουμε τον ακριβή αριθμό μελών για να μπορέσουμε να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία. Ξέχασα την κάρτα μου. Μπορείτε να λάβετε υπόψη τον τρόπο τον οποίο θα ψηφίσω. Πολύ ωραία το λαμβάνουμε, αλλά σηκώστε το χέρι σας καλά για να ξέρουμε αν ψηφίσατε υπέρ, κατά ή αν πέχετε από την ψηφοφορία. Λοιπόν, κάνουμε πρώτα απ' όλα το τεστ να δούμε αν δουλεύει σωστά το σύστημα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε όπω θέλετε. Δεν μετράει Ψήφο. Πρόκειται για τεστ. Πρόκειται για δοκιμή για να δούμε αν δουλεύει το σύστημα. Έληξε ψηφοφορία. 68. εφόσον ψήφισε η συνάδελφο υπέρ. Πολύ ωραία λοιπόν. Τώρα αρχίζει η πραγματική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εβδομηντα επτα υπέρ Δύο κατά και 22 εποχέ. Εγκρίνεται λοιπόν αυτή η απόφαση. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Λείτε η συνεδρίαση και σας ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Συνάδελφοι της Ήτρε, παρακαλώ να παραμείνετε στην αίθουσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της Επιτροπής Μεταφορών και την Πρόεδρο βεβαίως. Good morning once again. Uh, we start our uh, committee meeting of... Καλημέρα και πάλι. Ξαναρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα είναι η έγκριση μερίσης διάταξης. Έχουμε μπροστά μας το σχέδιο μερίσης διάταξης. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρώ ότι εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Σήμερα και πάλι είμαστε συνδεδεμένοι στο ίντερνετ. Έχουμε διερμηνία σε 22 γλώσσες. Η αποφάσεις των συντονιστών της 12 η Νοεμβρίου σας στάλησαν στις 26 Νοεμβρίου με email. Κάτι άλλο σημαντικό. Η απογευματινή συνεδρία της 5ης Δεκεμβρίου έχει καταρριχθεί. Πρώτα απ' όλα. Εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης 11 και 12 Νοεμβρίου Εάν συμφωνείτε, θεωρώ ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Περνούμε γρήγορα στο επόμενο θέμα. Ενημέρωση σχετικά με τι τρέχουσε διοργανικέ διαπραγματεύσει, σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλε ουσιώδει παραμέτρου. Η συγγήτρια από το ΕΛΚ, η κυρία Βερκούναν. Θέλω να σα πω ότι ο δεύτερος και τελευταίος διάλογος μεταξύ των τριών οργάνων έλαβε χώρα στις 13 Νοεμβρίου. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Βιρκούνεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Όπω είπε ο πρόεδρος, η δεύτερη συνεδρίαση του Τριμμένου Διαλόγου στις 15 Νοεμβρίου έφτασε σε μια προσωρινή συμφωνία. Θέλω να συγχαρώ, να ευχαριστήσω μάλλον τους κοιόδη ηγητέ, τους βοηθου τη γραμματεία, όλο τον κόσμο ο οποίος ε, έκανε πολύ καλή δουλειά. Τι θα γίνει τώρα με αυτές, με, ε, ε, με τη σήμανση, η σήμανση επικαιροποιήθηκε, μεγάλωσε. Ε, έχουμε το πικτόραμα του πάγου που είναι σημαντικό για τις βόρειες χώρες και ε, θα εφαρμόζεται η καινούργια ασήμανση και για λεωφορεία και για πούλμαν που δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή. Η, το βασικότερο θέμα που συζητήθηκε αφορούσε το, τα μικροπλαστικά ε, και τον χρόνο ζωής εκφρασμένο σε χιλιόμετρα. Ε, η έκτριψη δημιουργεί μικροπλαστικά και γι' αυτό το λόγο θα η Κομισιόν θα προτείνει ε, τρόπο μέτρησης μέσω μιας κατεξοδότησης πράξης όταν διαθέτουμε τις κατάλληλες μεθόδους. Ε, οπότε και η έκτριψη και η διάρκεια ζωής θα εμφανίζονται στις ετικέτες, στην σήμανση. Η, μόλις διαθέτουμε τις κατάλληλες μεθόδους μέτρησης θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε και την βιωσιμότητα ενός τέτοιου μέτρου ε, πάντως ε, ε, θα πρέπει να περιμένουμε να έχουμε τα οριστικά τέσσερις οριστικές μεθόδους δοκιμής. Αυτά θα ρυθμιστούν με πράξεις κατεξιοδότηση από την Κομισιόν. Ε, το θέμα ε, της ε, πρόσφυσης, ε, της αντίστασης και του θορύβου θα ρυθμιστούν με την συνήθη νομοθετική διαδικασία όταν στο μέλλον χρειαστεί να αλλάξουν οι παράμετροι. Θα χρειαστεί δηλαδή καινούριο νομοθετικό κείμενο. 1η Ιουνίου 2025 είναι η ημερομηνία εφαρμογής. Ε, ενώ η ε, θέση σε ισχύ γίνεται από το 2021, 1η Μαΐου του 2021. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεισέφεραν σε αυτή τη διαδικασία. Πρόεδρος, συγχαρητήρια σε εσά, στους και ηγητές. Θέλω να περάσουμε στην ψηφοφορία κατευθείαν. Πρώτα θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Δοκιμαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίστε ό,τι θέλετε, υπέρ, κατά, αποχή. It's okay, It's okay. Ωραία είμαστε. Περνάμε τώρα στην κανονική ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Everybody voted. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία, λίγη ψηφοφορία. Strong. Ισχυρή πλειοψηφία, συντριπτική πλειοψηφία υπέρ. Με δύο εποχές. Συγχαρητήρια μία ακόμα φορά και καλή τύχη για το μέλλον. Περνάμε στο σημείο 7. Ε, ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ζων Ερικ Πακέ, Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας. Η ανταλλαγή απόψεων θα αφορά τις εταιρικέ σχέσεις και τις αποστολές στο πλαίσιο του προγράμματος ε, Horizon Ευρώπη. Παρακαλώ πολύ όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, ας ε, το κάνετε όσο πιο ήσυχα γίνεται. ορίζω, λοιπόν το Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Πακέ, ο οποίος μας επισκέφθηκε και το Σεπτέμβρη. Η παρουσία του σήμερα αποδεικνύει μια φορά ακόμα φορά το ενδιαφέρον που δείχνει η Επιτροπή μας στο στρατηγικό σχεδιασμό του προγράμματος Horizon Europe, καθώς επίσης και την βούληση της Κομισιόν να είναι σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο συχνά το απαιτούν οι περιστάσεις. Σήμερα θα μάθουμε περισσότερα για την εξέλιξη του στρατηγικού σχεδιασμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αποστολέ και τις εταιρικές σχέσεις. Ε, και ό,τι καινούριο έχουμε σε σχέση με την τελευταία μα συνεδρίαση. Πιο συγκεκριμένα, τι λεπτομέρειε για τα επόμενα βήματα του στρατηγικού σχεδιασμού και τη ε, διαδικασία του. Επίση, ε, λεπτομέρειε για το πώ επιλέγονται οι εταιρικέ σχέσει συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών σχέσεων μεταξύ κρατικών φορέων, PPP δηλαδή, και των πρωτο... κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλειών. Και επίση πώς ορίζονται οι αποστολές ε, σε, με συγκεκριμένα μέτρα, ε, συγκεκριμένα λόγια. Ε, μία ώρα και 25 λεπτά θα αφιερώσουμε σε αυτό το θέμα. Θα δώσω το λόγο καταρχήν στον κύριο Πακέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Συγχαρητήρια και από εμένα για την εκλογή σας. Αναμένω την συνεργασία μας και σας ευχαριστώ για την δυνατότητα μου δίνετε να μιλήσω στην Επιτροπή σας ε, εξ ονόματος της ε, Επιτρόπου της κυρίας ε, Γκάμπριελ καθώς είχε δεσμευτεί κατά τη διάρκεια της ακροάσης για το ότι θα ενημερώνει Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας για τις εξελίξεις του πρόγραμμα Ορίζοντας για την Ευρώπη. Μάλιστα είχα την τιμή να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας ε, αρχές ε, Σεπτεμβρίου για να σας ενημερώσω για τα τρέχοντα και θα προσπαθήσω τώρα να αναφερθώ στις ε, κύριες εξελίξεις έκτοτε. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα και μετά να μένω τις ερωτήσεις για τα διάφορα στοιχεία των, της προετοιμασίας αυτής. Το πρώτο το οποίο έχω να πω είναι ότι είχαμε μια πολύ εντυπωσιακή συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην Ευρώπη μέσω της ε, δημοσίας ε, διαβούλευσης. Ε, τα κάλυψα αυτά όταν συναντηθήκαμε. Έκλεισε 4 Οκτωβρίου. Λάβαμε 6.806 απαντήσεις στην δημόσια διαβούλευση. Μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν από τους εταίρους ανά την Ευρώπη πως η διαδικασία αυτή έχει αντίκτυπο στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος. Μετά είχαμε τρεις μέρες ε, εντατικής και άμεσης ε, ανάδρασης ε, και συνεννόηση μεταξύ των κοινωτικών υπαλλήλων και των εθνικών διοικήσεων και των ενδιαφερομένων και χαίρομαι για το ότι και πολλοί βουλευτές ήταν παρόντες στις μέρες έρευνας και καινοτομίας και συνεισέφεραν στις συζητήσεις. Η διαδικασία αυτή λοιπόν από κοινού σχεδιασμού του προγράμματος Ορίζοντας για την Ευρώπη υλοποιήθηκε κατά τις τρεις αυτές ημέρες και νομίζω ότι ο αντίκτυπος ήταν πάρα πολύ ε, ουσιαστικός. Αυτό το οποίο έκανε μετά η Κομισιόν είναι να επικαιροποιήσει το έργο της και είχαμε στο τέλος Οκτωβρίου ένα πιο ενημερωμένο έγγραφο, το οποίο βεβαίως δώσαμε στη γραμματεία της Επιτροπής σας. Και βεβαίως υπάρχει άλλος επιπλέον γύρος πιο στοχευμένων σχολείων και βεβαίως πάντα είμαστε στην διάθεση του κοινού για να απαντήσουμε λάβαμε και κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις που εν ολίγης επιβεβαιώνουν τις επιλογές ε, ε, τον αντίκτυπο που ανέφερα κάτι το οποίο βεβαίως ε, θα καθοδηγεί και τη νέα επιτροπή της κυρίας Ούρσουλα Φόντερ Λάιν και στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων και με την γραμματεία της Επιτροπής Ήτρε και με τους βουλευτές ε, είδαμε κάποιες σκηνές ε, προκλήσεις στα διάφορε, στις διάφορες δέσμες, παραδείγματος χάρη πράσινη πληροφορική, κάποια άλλα επιπρόσθετα μέτρα τα οποία προέκυψαν ε, για να εστιάσουμε περισσότερο στα ανοιχτά επιστημονικά δεδομένα και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δούμε τον πιθανό αντίκτυπο των συνεργειών μεταξύ του προγράμματος συνδέοντας την Ευρώπη και των άλλων στοιχείων του μελλοντικού ευρωπαϊκού προπολογισμού. Τώρα, έχουμε ένα σχεδόν σταθερό εγγραφό το οποίο θα είναι διαθέσιμο πρόσεχώς Και βεβαίως ε, με βάση αυτό θα συνεργαστούμε με το προσωπικό για να καταρτήσουμε τον πιο λεπτομερή στρατηγικό σχεδιασμό και αυτό βεβαίως ε, θα πρέπει να λάβει υπόψη ε, και την δουλειά που γίνεται στο πλαίσιο του μελλοντικού ΠΔΠ γιατί θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να οριστικοποιήσουμε τις προετοιμασίες χωρίς να γνωρίζουμε τον τίτλο του προγράμματος, τον αριθμό μου συγχωρείτε, το ύψος και την ε, κατανομή του βεβαίω την οποία θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα θεσμικά όργανα. Στο πλαίσιο αυτό, να πω δύο λόγια για κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία που νομίζω σας ενδιαφέρουν. Το πρώτο είναι οι αποστολές και το δεύτερο οι συνεργασίες για τις αποστολές. Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι το Συμβούλιο Αποστολών που συστάθηκε το καλοκαίρι για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για τον καρκίνο, για το ύδατα, ωκεανούς, ποταμούς λοιπά Για τις πόλεις και το έδαφος και τα τρόφιμα. Όλες αυτές οι ομάδες έχουν συνεδριάσει τουλάχιστον δύο φορές Μάλιστα η Επιτροπή για τις Πόλεις ήδη τέσσερις φορές και αναμένουμε ότι ε, θα μπορέσουν να επανέλθουν στην Κομισιόν αλλά να είναι σε επαφή και με το Κοινοβούλιο για τις ε, συμβουλές τους για το ποιος θα είναι ο στόχος. Λοιπόν, έχουμε φτάσει τώρα στο επίπεδο των ε, περιοχών ε, και βέβαια αναμένουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των αποστολών αυτών. Στη ε, πλαίσιο αυτής της διαδικασίας συνεργαζόμαστε με τα συμβούλια αυτά και τις εθνικές διοικήσεις και η Μαρία Γκαμπριέλ νομίζω ήλπιζε για μια μεγαλύτερη εμπλοκή των βουλευτών για να μπορέσουμε να έχουμε ε, συμμετέχοντες σε αυτές τις αποστολές, ε, δηλαδή επιστήμονες, πανεπιστήμια, αλλά και ε, τοπικούς φορείς, πολίτες και τα σχετικά. Όπως είπε ο Κάρλος Μάγιος, το νόημα είναι ακριβώς να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε την φαντασία της ευρωπαϊκής κοινή γνώμης, να βρεθεί δηλαδή ο κατάλληλος τρόπος να είμαστε σε επαφή με τους Ευρωπαίους πολίτες, να φανεί αυτό, να ακούσουμε τα όσα έχουν να πει και να σχεδιάσουμε μαζί τους ε, τις αποστολές. Νομίζω ότι θα έχουμε έτσι μια σημαντική συνεισφορά σε αυτό το θέμα, μια διαβούλευση δηλαδή, η οποία αν είναι επιτυχής ε, θα βοηθήσει στην επιτυχία των αποστολών. Έτσι λοιπόν έχει συζήτηση αυτή τη στιγμή το πώς θα μπορέσουν να ταξιδέψουν οι αποστόλες αυτές σε όλα τα κρατημέλη και να είναι σε επαφή με τους πολίτες. Οπότε ενδιαφέρον οι προτάσεις από τους ε, βουλευτές ε, ε, είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Επίσης η κυρία Γκαμπριέλ είπε ότι θα ζητήσει κάθε να είναι από αυτά τα Συμβουλία Αποστολής να ορίσει κάποιον σύνδεσμο με την Επιτροπή σας. Αυτό έχει ε, σχεδόν γίνει τώρα και η Κομισιόν ε, θα σας απευθύνει μια επιστολή με τα ονόματα για να μπορέσετε να ξεκινήσετε την συνεργασία. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι η Επιτροπή σχεδιάζει μια ακρόαση και βεβαίω ε, αν μπορούμε να Σα στηρίξουμε σε αυτό. Ευχαριστώ να το κάνουμε. Μία τελευταία λέξη για τις ε, συνεργασίε. Εδώ πέρα επίσης είχαμε κάποιες εξελίξεις ε, στο θέμα του προσανατολισμού του στρατηγικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα έχουμε τώρα ε, λαμβάνοντας υπόψη και τις συζητήσεις εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε 48 εταιρικές σχέσεις για τις οποίες συνεχίζεται το προπαρασκευαστικό έργο. 13 ε, διοργανικές ε, τέτοιες ε, θεσμικές σχέσεις οι οποίες αναλύονται εντός της Κομισιόν η οποία θα τις εφαρμόσει κιόλας. Νομίζω ότι αυτό το είχε ξεκαθαρίσει και η Επίτροπος και θα το συζητήσουμε τον Σεπτέμβριο Δηλαδή έχουμε δει το προς που θα κινηθούν αυτές οι συνεργασίες, αλλά πρέπει να επιβεβαιώσει και η ανάλυση ή όχι το εάν αυτή η πολύ προχωρημένη μορφή ε, θεσμικής ε, συνεργασίας έχει κάποια σχέση. Και βεβαίως το αν ε, θα είναι πιο ουσιαστικό από την πλευρά της συγχρηματοδότησης. Και βεβαίως ε, τώρα συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς της Εθνικής Διοίκησης και οργανώσεις έρευνας ε, για να προετοιμάσουμε το έδαφος για την μελλοντική εφαρμογή και νομίζω αξιοσημείωτο είναι το ότι έχουμε προσθέσει τέσσερις επιπλέον ε, συνεργασίες ε, στο έγγραφο που είχατε δει πριν από το καλοκαίρι οι οποίες ε, καλύπτουν την υγεία και την αντίσταση στα μικρόβια, έξυπνες πόλεις και κοινότητες και βεβαίω αυτό σχετίζεται και με την αποστολή για τις πόλεις και επίσης υδατικές και γεωλογικές υπηρεσίες Έχουμε λοιπόν αυξή από τις 44 στις 48 συνεργασίες επί των οποίων εργάζονται οι υπηρεσίες κομισιών και βεβαίως το έργο υλοποιείται στο επίπεδο των νομοθετικών προτάσεων. Λοιπόν, εάν συμφωνείτε θα σταματήσω εδώ και είμαι στην διάθεσή σας για να απαντήσω για τις άλλες πτυχές ε, του ορίζοντα Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εξηγήσεις σας και για την ε, δεκτικότητά σας. Ε, δηλώσατε ότι θέλετε να συναστείτε με το Κοινοβούλιο. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα στον κόσμο σε αυτού του είδους το Horizon Europe. Ε, έχουμε κάνει πολλά βήματα θετικά, έχουμε και βελτιώσει βέβαια να γίνουν. Θα δώσω το λόγο στους συντονιστές και μετά θα δώσω το λόγο σε άλλους ε, βουλευτές που τον θέλουν. Θα ξεκινήσω με τον συντονιστή του ΕΛΚ, ε, που είναι και εισηγητής για το πρόγραμμα Horizon Europe. Θα ξεκινήσω με κάποια διαρθρωτικά θέματα, λέει ο κύριος Έλλερ. Η διαδικασία διαβουλεύση είναι αρκετά ανοιχτή, αλλά και έχουμε εντοπίσει κάποιες διαφορές ανάμεσα στο, προ, στο ε, έγγραφο προσανατολισμού και στην μερική συμφωνία. Για παράδειγμα, το επωνομαζόμενο climate kick δεν αναφέρεται Ε, Επίση το CCI δεν αναφέρεται στο κλάστερ 2. Ε, η ισορροπία ανάμεσα στις στρατιωτικές και πολιτικές πτυχές έρευνα. θα έπρεπε επίσης να, να αναφέρεται στην πολιτική συμφωνία για το Horizon Europe στα συγκεκριμένα προγράμματα, ιδιαίτερα στην εισαγωγή. Είναι τεχνικής φύσεως βέβαια, αλλά ε, έχει πολλή ουσία αυτό που λέω. Μετά, πώς οι αποστολές θα συνδέονται με προηγούμενες στρατηγικές και πρωτοβουλίες όπως η πρωτοβουλία για τις ευφύς πόλεις. Δεύτερον, τα έξι προεπιλεγμένα σχέδια πώς θα συνδέονται με τις αποστολές. Ε, 1,5 εκατομμύριο λαμβάνουν και δεν ξέρουμε πού θα ενταχθούν. Μετά, η συνέπεια με τον οικονομικό κανονισμό. Ε, υπάρχουν κάποιες καθαρές γραμμέ οι οποίες δημιουργούν σύγχυση για τις ε, εταιρικές σχέσεις, διότι ε, προσπαθούν να αποτρέψουν ε, τα ε, κράτη να γίνουν με τμήματα ιδιωτικών εταιρικών σχέσεων. Η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντο για προτάσει, υποβολή προτάσεων, θα πρέπει να είναι ανοιχτή όμω και στα κράτη-μέλη και σε μη Και σε μη φορού. Οπότε δεν είναι σαφές το πόσο θα εξασφαλιστεί η ισορροπία ανάμεσα στους κρατικούς και τους δημόσιους φορείς και τους ιδιωτικούς φορείς. Μετά ένα θέμα διακυβέρνησης. Πώς εντάσσουμε τις πρόσφατες φιλοδοξίε για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, 55%. Δηλαδή Σε ορισμένες σχέσεις, τις οποίες εξετάζουμε, για παράδειγμα, ε, οι εκπομπέ από την αεροπορία είναι τρεις φορές περισσότερες από τις ε, μειώσεις που γίνονται. Ε, οπότε πώς θα πετύχουμε το στόχο του 55%. Δηλαδή έχουμε καινούριε φιλοδοξίες από την Κομισιόν, από την άλλη μεριά έχουμε μια, ένα στρατηγικό σχεδιασμό ο οποίος ακόμα κινείται στα παλιά δεδομένα. Μια άλλη τεχνική ερώτηση. Έχουμε ένα κατάλογο 44 εταιρικών σχέσεων, μόνο 13 όμως έχουν μελέτες επιπτώσεων. Ποια θα είναι η μεθοδολογία θα γίνουν ε, τέτοιου είδου μελέτες μόνο για κάποια μερικέ από τι εταιρικέ σχέσει κλειδί, Όπω για παράδειγμα το καθαρό υδρογόνο. Μετά, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο στρατηγικό σχεδιασμό και τις φιλοδοξίε σε ό,τι αφορά τα προγράμματα εργασία αργότερα. Γίνεται ένα μείγμα, μάλλον αναμειγνύονται, συγχέονται αυτά τα δύο. Τελευταία μου ερώτηση Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το, ε, ε, το, ευρωπαϊκό, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας ε, αποκλείεται κατά κάποιο τρόπο εν μέρη. Θα έπρεπε να καταλάβουμε καλύτερα πώς συνδέονται που συνδέεται η εργασία του ποια, ποιος είναι ο ρόλος του. Ε, ζητώ συγγνώμη που μπαίνω σε λεπτομέρειες, αλλά θα προκύψουν αυτά τα θέματα. Οι συντονιστές αποφάσισαν να γίνει μια ακρόαση με τι επιτροπή Ήτρες το Φεβρουάριο, στι 18 Φεβρουαρίου, οπότε θα ήθελα η Κομισιόν να συμμετάσχει. Thank you very much, uh, Mr. I hope you know... Πρόεδρος, ελπίζω ο κ. Πακέ να σημείωσε τι ερωτήσει όλες. Ο κ. Ντανίκα, συντονιστής των σοσιαλιστών, αλλά και εισηγητής για το πλαίσιο του Ορίζων Ευρώπη. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας. Και ελπίζω να συνεχίσετε την ε, παράδοση του κ. Μπούζεκ σε αυτή την Επιτροπή. Θα πρέπει να υπερασπιστείτε τις αρμοδιότητές μας, να προασπίσετε τις αρμοδιότητές μας και να μας βοηθήσετε να εργαστούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμείς θα σας βοηθήσουμε. Να καλωσορίσω τον κύριο Πακέ. έχω περάσει μερόνυχτα μαζί τους στον τριμερή διάλογο για να βρούμε μια λύση την οποία στηρίζουμε και πρέπει να γίνει σεβαστή. Η πολιτική συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντική, μας προσιάσατε αρκετές λεπτομέρειες και η κυρία Γκαμπρίελ και εσείς ο ίδιος δείχνετε ανοιχτή έναν των θέσεων του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι πολύ καλό. Και ελπίζω να συνεργαστούμε. Αυτό που θα πω νομίζω ότι το συμμερίζονται και άλλοι σκιοδησηγητές. Το πρόγραμμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Κάναμε μια πρόταση την οποία στήριξε η Φιλανδική Προεδρία. Αλλά υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τα οποία διαφωνούν. Οι μειώσεις και οι περικοπές που προτείνουν είναι απαράδεκτες. το ποσό το οποίο το κοινο, που πρότεινε το Κοινοβουλίο βασίστηκε στην ανάγκη να επιτευχθούν οι στόχοι. Πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας τους στόχους του, της Νέας Πράσινης Συμφωνίας και της μείωσης ε, της χρήσης του άνθρακα, αν γνωρίζουμε ότι με την τεχνολογία που διαθέτουμε σήμερα τα πράγματα είναι ή πολύ δύσκολα ή αδύνατα. Επίσης, κάποια κράτη-μέλη ε, θέλουν μείωση των κονδυλίων για την έρευνα. Πώς θα πετύχουμε τη μείωση της χρήσης του άνθρακα χωρίς επαρκή χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, αποθήκευση ενέργειας. Το 99% ε, της αποθήκευσης γίνεται με τεχνολογίες που ε, μετρούν 50 χρόνια ζωής. Έχουμε χάσει το τρένο της ε, έρευνας στις ε, μπαταρίες στις ισορρευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Χρειαζόμαστε επαρκή χρηματοδότηση για να ξαναβρούμε τη θέση μας. Αυτό είναι σημαντικό για όλους τους παρα... οικονομικούς ε, φορείς και τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να μειώσουμε κατά 50-55% τα αέρια θερμοκηπίου, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Αυτή είναι, αυτός είναι ο καινούριο στόχος. Συμφωνούμε και στηρίζουμε αυτή την επιλογή, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση. Αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να, να ηγηθούμε της ε, παγκόσμια προσπάθειας εναντίον τη κλιματική αλλαγή. Αν δεν έχουμε ούτε επαρκή χρηματοδότηση, ούτε επαρκή ε, προτεραιότητε, ε, δεν θα πετύχουμε το στόχο μας. Τώρα, οι προτάσεις για τις εταιρικέ σχέσεις θα δημοσιευτούν πριν να υιοθετηθεί το ε, πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό είναι μια φήμη ενδεχομένω. Θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε να το διαψεύσετε. Έχουμε μια πρόταση πλαίσιο για όλε τι εταιρικέ σχέσει. Και αν το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίση αν το Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία θα συνεισφέρει Και η τελευταία μου ερώτηση είναι η Ποια σχέδια είναι τα, αυτά που είναι πιο προχωρημένα για δημιουργία εταιρικών σχέσεων. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που δείχνετε διάθεση συνεργασίας και ελπίζω ότι θα προκύψει κάτι καλό γιατί εξαρτώνται πολλά για, στο μέλλον ε, από την ε, δική μας ε, στάση αυτή τη στιγμή. Σε e. ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Επιτροπής μας. Από την κυρία Τζαβάραβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια και αναμένω την ε, συνεργασία μας τα επόμενα χρόνια. Κύριε Βακέ, σε ένα γενικό επίπεδο, α, ε, ανησυχώ ε, από τα όσα ακούμε από το Συμβούλιο σχέση με το ΠΔΠ και τον ορίζοντα της Ευρώπης. Βεβαίως μιλάμε για μεγάλα ποσά, αλλά Δεδομένη της προσθέμενης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το ότι μιλάμε για το ότι η έρευνα και η καινοτομία θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και το ότι έχει μείνει πίσω η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αναρωτιέμαι γιατί δεν ε, δίνουμε περισσότερα λεφτά σε αυτό το πρόγραμμα. Τι κάνουμε λάθο, ποιο είναι το αφήγημα που πρέπει να φτιάξουμε για να τα πάμε καλύτερα. Ναι, επί του οποίου θα μπορούσαμε να εργαστούμε καλύτερα ως ε, Κομισιόν και, Συμβούλιο για να πει, Κομισιόν και Κοινοβούλιο για να πείσουμε το Συμβούλιο γιατί ζητήσαμε 150 δισεκατομμύρια αλλά ε, δεν έχουμε ακόμα πλησιάσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί η προηγούμενη Κομισιόν. Δεν ξέρω αν ε, συμφωνείτε. Έχω και μια συγκεκριμένη ερώτηση για τα μέσα του προγράμματος Horizon. Η Κομισιόν έχει ένα αρκετά καλό κείμενο στο άρθρο 11 του κανονισμού και αφορά την συνέργεια και δεν έχει συζητηθεί ακόμα στις τριμερεί διαπραγματεύσεις. Το άρθρο λοιπόν λέει το εξής. η ε, Ευρώπη θα πρέπει να εφαρμοστεί σε συνέργεια με άλλα προγράμματα χρηματοδότησης επιδιώκοντας τη μέγιστη διοικητική απλοποίηση. Ένας μη εξαντλητικό ε, κατάλογος συνέργειας με άλλα προγράμματα περιλαμβάνεται στο παράρτημα 4 οι ενιαίοι κανόνες θα ισχύσουν για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις. Οπότε, εγώ συνεργάζομαι με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θεωρώ ότι πρέπει να εμπλακούν ακόμη περισσότερο στο πρόγραμμα. Θα διασφαλίσετε ότι στο μέτρο του δυνατού οι ενιαίοι κανόνες θα ισχύσουν στις σχετικές ε, δράσεις. Ε, είτε μιλάμε για ε, σχέση συνεργασίας ή ε, καινοτομίας γιατί πραγματικά είναι αποκαρδιωτικό όταν μιλάμε για μικρόμεσαίες επιχειρήσεις και μετά από τον πρώτο γύρο που καταναλώνουν χρήμα και χρόνο παρατηρούν ότι έχει τελείως διαφορετικούς κανόνες ο στόχος για τον οποίο έχουν ζητήσει χρηματοδότηση. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν στο πεδίο της συνέργειας και της απλοποίησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τους πράσινους η κυρία Τζίνα Ντάουντινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πακέ, σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας και για το ότι δέχεστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Εάν είναι λοιπόν, αν πρόκειται να κάνει τη διαφορά η ευρωπαϊκή έρευνα, θα πρέπει να καθοδηγείται από τις προτεραιότητες της κοινωνίας. Γι' αυτό έχει σημασία να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι στη διαμόρφωση των προγραμμάτων για να αντιμετωπίζονται τα πιεστικά προβλήματα, η κλιματική αλλαγή, η πράσινη μετάβαση και η υγεία όμως. Εάν η εμπλοκή της κοινωνίας ε, μειωθεί, ε, η διαδικασία αυτή του αποκοινού σχεδιασμού μπορεί να αποδειχθεί και αντιπαραγωγική. Γι' αυτό ε, οι πρόσφατοι αριθμοί από τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού μας ανησυχούν από 1.549 συμμετοχές, μόλις 95 ήταν από μήκαιο και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Και ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις ε, έδωσαν 542 απαντήσεις. Φοβούμε λοιπόν ότι υπάρχει ο κίνδυνος εδώ να κυριαρχήσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Τώρα η συμμετοχή θα πρέπει να εστιαστεί σε πιο Συγκεκριμένε προτεραιότητε, Πολλές εκθέσει το λένε αυτό και αμφισβήτησαν το εάν οι προτεραιότητε αυτές έχουν πραγματικά ωφέλη για τους ε, πολίτες. Και αυτό φαίνεται ιδιαίτερο στα κοινά εγχειρήματα, ναι, καθώς η ερευνητική του ατζέντα κυρίω ε, αφορά τις βιομηχανίε. Με τόσο χαμηλή συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών στον τελευταίο γύρο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού, θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτα, πώς σκοπεύετε να αυξήσετε την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού και στην εφαρμογή του ορίζοντα για την Ευρώπη. Και δεύτερον, δεδομένου του ότι η Κομισιόν σκοπεύει να ανανεώσει τις ε, εταιρικές σχέσεις του κοινού εγχειρήματο, πώς σκοπεύετε να υπερασπιστείτε το δημόσιο συμφέρον και να χρηματοδοτείτε πράγματα τα οποία όντως θα ωφελήσουν την κοινωνία και θα είναι προσβάσιμα σε όλους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ για τις ερωτήσεις σας. Για την ομάδα ID, ο κύριος Μποργία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας ε, κύριε Πακέ για την εισαγωγή σας μία σύντομη ερώτηση που σχετίζεται και με αυτά τα οποία είπαν κάποιοι προλαλήσαντες. Δεδομένου του ότι με το Horizon 2020 οι εταίροι ε, δεν υπάρχει μάλλον η δυσκολία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση γιατί δεν ρισκάρουν όλοι μια συμμετοχή σε μια τέτοια συνεργασία και δεδομένου του ότι όταν υλοποιούνται αυτές οι συνεργασίες είδαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι μεγαλύτεροι εταίροι έχουν υποβιβάσει τους μικρότερους σε έναν πιο ε, περιθωριακό ρόλο θα ήθελα να γνωρίζω εάν και πώς σκέφτεστε στο Horizon Europe ε, οι συνεργασίες αυτές ε, θα μπορούσαν να ε, πιθανώς να αναδείξουν περισσότερο τον ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς ε, βεβαίως υπάρχουν αυτές οι διαφορές μεγέθους μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Για το ECR τώρα, ο κύριος Κρασνοντέρσκι. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ. Να... Πω το εξής. Μιλούμε για διάφορες εταιρικέ σχέσεις και συμπράξεις και το ερώτημά μου σε σχέση με το θέμα αυτό αφορά τις αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο κατάλογο. Έχει γίνει ποιοτικέ αλλαχές. Έχουν γίνει προσπάθειες για να γίνει πιο ενδυτική η έρευνα έτσι όπως το προτείνει η Κομίσια. Είχαμε έναν ε, πιο εκτενή κατάλογο. Μπορείτε να μου πείτε κάποια από τα θέματα που πραγματεύονται αυτού του είδους οι έρευνες. Εγώ μίλησα με κάποιους ενδεχόμενους υποψηφίους οι οποίοι έχουν κάποια ερωτηματικά σε σχέση με το τι μπορεί κάποια, με, πώς μπορεί να το εντάξει όλο αυτό το εγχείρημα κάθε χώρα θα υπάρχει ε, κάποια συμμετοχή των διαρθρωτικών ταμείων, μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε αυτό να θεωρηθεί ε, σαν ε, συμμετοχή μιας χώρας χωρίς να θεωρηθούν ότι δίδονται κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όσον αφορά την χρηματοδότηση, τις συμπράξεις αυτές, πώς θα γίνει ακριβώς η χρηματοδότηση. Θα υπάρξουν σχέδια συνεργασίας, μεταφορά κονδυλίων στα πλαίσια του Horizon Europe. Νομίζω ότι τα σχέδια και τα προγράμματα συνεργασίας θα πρέπει να αποτελούν το κύριο σώμα. Προβλέπετε λοιπόν τέτοιου είδους μεταφορές κονδυλίων. Επίσης, η ποιότητα, όπως είπαμε, της έρευνας, η χρηματοδότηση και η κατάλογοι, όπως σας είπα, θεωρώ ότι είναι σημαντικά θέματα, γι' αυτό θα ήθελα εξηγήσει εκ μέρους σας. Σας ευχαριστούμε. Τελευταία, αλλά η κυρία Μαρίζα Ματία, τελευταία λόγια λιγότερο σημαντή στην. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για την εκλογή σας Πρόεδρε. Κύριε Πακέ, σας καλωσορίζω και πάλι στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι μας παρουσιάσατε πολλά στοιχεία περισσότερο από θέματα γενικά στρατηγικής και μιλήσατε και για τις συμπράξεις. Ξέρετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο την ιδέα να έχουμε νέα μέσα την ε, θεωρήσαμε πολύ θετική από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι έτσι μπορούμε να αναπτύξουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ερευνών και οργανωτικής και διαστορωτικής Πλευρά επίσης αυτό είναι σημαντικό. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή μας σε κάποια ευάλωτα σημεία και σε κάποια προβλήματα και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να απορρέουν από αυτή την πρόσθεση νέων μέσων εάν δεν γίνουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Ήδη έχουν τεθεί κάποια ερωτήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την ύπαρξη προβλημάτων και πρέπει να τα αποφύγουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τώρα, υπάρχει πρώτα απ' το πρόβλημα των κονδυλίων από τον προϋπολογισμό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν επιλογές. Υπάρχει ήδη καθορισμένη ε, σχέση, ε, απόφαση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν γίνουν αυτές οι επιλογές για να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε. Δεύτερο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου το θέμα των ε, συνεργειών μεταξύ των διαφόρων μέσω χρηματοδότηση. Πάλι και αυτό θέλω διευκρίνηση. Και κατά την άποψή μου κάτι άλλο το οποίο επίσης είναι σημαντικό για μένα είναι συμπληρωματικότητα μεταξύ των νέων μέσων και των μέσων των ε, οργανισμών που υπάρχουν ήδη στα πλαίσια του Horizon Europe. Φερρυπίν. Το ΕΙΤ εντάχθηκε εδώ, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο, στο Horizon Europa. Αλλά στην παρουσίασή σας δεν το αναφέρατε συγκεκριμένα. Το θέμα του κλίματος επίσης αναφέρεται. Το AT ξέρουμε ότι είναι μέρος του στρατηγικού σχεδίου. Το να το έχουμε κάπου απανομένα μπορεί να είναι μία μορφή μη διευκρίνησης κάποιων μέσων. Και τι κινδυνεύουμε, να δημιουργήσουμε μέσα και μηχανισμούς που δεν θα μπορέσουν να εξελιχθούν κανονικά. Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε αυτό. Πώς βλέπετε εσείς τη συμπληρωματικότητα λοιπόν όλων αυτών των νέων μέσων, των εταιρικών σχέσεων, των αποστολών με αυτού που ήδη υπάρχουν και κυρίως να αναφερθώ στο EET δεδομένου ότι δεν το διευκρινίσατε κατά τη διάρκεια της παρέμβασής σας. Νομίζω ότι όταν θα διευκρινιστεί αυτή η συμπληρωματικότητα θα είμαστε πιο ήσυχοι, δεδομένου ότι θα μπορούσαμε, αν δεν έχουμε πλήρη περιγραφή και γνώση, να δημιουργήσουμε το κουτί της Πανδώρας, όταν το ανοίξουμε μπορεί να χάσουμε πολλά. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε με τις ερωτήσεις τα σχόλια των συντονιστών. Πολλές οι ερωτήσεις. Θα απαντήσει ο κ. Πακέ και μετά θα δώσω το λόγο σε 7 συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν για λιγότερο χρονικό διάστημα ο καθένας, αλλά εξίσου σημαντικά τα σχολεία τους φαντάζομαι. Ο κ. Πακέ έχει το λόγο. Πολλές οι ερωτήσεις, θα κάνω ό,τι μπορώ. Πολλές ερωτήσεις τις έχουμε και εμείς ε, στο μυαλό μας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά να συζητήσουμε όλα να συνεχίσουμε κιόλας συζήτηση αργότερα, αν μείνει κάτι αναπάντητο. Να ξεκινήσω με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Καινοτομίας, στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Ματίας, αλλά και ο κύριος Έλερ και άλλοι. Αποτελεί τμήμα του στρατηγικού σχεδιασμού όλης αυτής της διαδικασίας για πρώτη φορά. Ασφαλώς θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συνδεθούν, θα συνδεθούν οι αρεσίες του Ινστιτούτου με τις γενικότερες προτεραιότητες. Δεν ήξερα ότι το climate kick δεν έχει αναφερθεί. Πρέπει να αναφερθεί. Σωστό. Είναι εύκολο να το διορθώσουμε αυτό. Και αυτό φορά όλα τα kicks γιατί εντοπίζονται συγκεκριμένα στον κατάλογο των εταιρικών σχέσεων, των συνεργασιών. Και μάλιστα συζητούμε ήδη το μελλοντικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού, Τεχνολογικού Ιδρύματος, ε, Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Τεχνολογίας και Και μαζί με τον κανονισμό ε, συζητούμε και την ε, πρακτική εφαρμογή, το πρακτική, τον πρακτικό καθορισμό του προγράμματος εργασίας του Ινστιτούτου, το οποίο πρόγραμμα εργασίας θα συνδέεται άμεσα με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες του ορίζον Ευρώπη. Ας μην υπάρχει κανονός είδους αμφιβολία γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, εργαστούν για τους ίδιους σκοπούς. Έχουμε πλέον μία μόνο επίτροπο που καλύπτει όλα αυτά τα θέματα, οπότε είναι ευκολότερο να γίνει ο συντονισμός. Για τα ΦΕΤ, Ε, και τα προεπιλεχθέντα. Όσα ήδη υπάρχουν, ε, ε, όσες μιλάμε για τις μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες, όσες ήδη έχουν ξεκινήσει θα συνεχιστούν. Προσπαθούμε να καλύψουμε ε, τις καινούργιες και να δούμε ποια είναι η σχέση τους με ήδη υπάρχουσες ε, εταιρικές σχέσεις για να δούμε πώς ακριβώς θα συνδυαστούν με τις παλαιότερες. Οπότε τις μελλοντικές και αναδέωμες τεχνολογίες τις έχουμε υπόψη μας και οι έξι που έχουν προεπιλεγεί θα λάβουν ε, μεγάλη σημασία, θα αποκτήσουν μεγάλη σημασία για το μέλλον. Τώρα, δεν βλέπω τις ε, αντιφάσεις με τον οικονομικό κανονισμό. Θα πω όμως στους δικηγόρου να το ξανακοιτάξουν. Υπάρχει περίπτωση. Είναι σαφές πάντως ότι το να προωθήσουμε περισσότερες επενδύσεις στις εταιρικές σχέσεις είναι απολύτως απαραίτητο Αν θέλουμε να δούμε ε, εταιρικές σχέσεις όπως για παράδειγμα για την αεροπορία, την πολιτική αεροπορία, ε, όλα αυτά, όλα αυτά θα γίνουν εν μέρη και με κρατική χρηματοδότηση βέβαια, αλλά σίγουρα όχι μόνο με κρατική χρηματοδότηση, χρειαζόμαστε και ιδιωτικές επενδύσεις Κατανοώ πως είναι περίπλοκο. Είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε την διαφάνεια των επενδύσεων από ιδιωτικού ε, φορεί και να εξασφαλίσουμε μάλιστα μετά ότι ο φορέα θα εφαρμόσει αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί. Το σκεφτόμαστε. Εξετάζουμε και το θέμα των μελετών αντικτύπου Ποιος ρώτησε για το αν θα υπάρχει μία μόνο νομική πρόταση ενιαία για όλες τις ε, εταιρικέ σχέσεις. Δεν το έχουμε αποφασίσει αυτό. Από ό,τι φαίνεται όμως υπάρχουν πολλές διατάξεις, πολλές ρήτρε που θα είναι ίδιες για όλες τις εταιρικέ σχέσεις. Για παράδειγμα, ο αντίκτυπος στην κοινωνία. Οπότε θα θέλαμε πράγματι όλες τις εταιρικές σχέσεις να τις ε, ε, συντονίσουμε, να τις ενοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πολύ κατακαιρματισμένες, κάθε μία δουλεύει προς τη δική της κατεύθυνση. Ε, οπότε, αν είχαμε μία, ένα ενιαίο νομικό κείμενο που θα είχε τις ίδιες λίγος πολύ ρήτρε, θα, ε, θα ήταν χρήσιμο. Θα το, θα το αναλύσουμε όμως περαιτέρω αυτό. Επίσης, θα βρούμε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να εξασφαλίσουμε περισσότερη χρηματοδότηση από τους διάφορους κλάδους, τον ιδιωτικό τομέα. Ε, 13 ε, μελέτες επιπτώσεων έχουν ολοκληρωθεί, όμως θα χρειαστούν και οι υπόλοιπε. Για τις υπόλοιπε δηλαδή εταιρικές σχέσεις. Ε, μιλήσατε για τις εταιρικές κλειδί, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς η εφαρμογή θα επιτρέψει και μια αποτελεσματική παραγωγή, βιομηχανική παραγωγή στον αντίστοιχο κλάδο. Οπότε θα πρέπει και ο ίδιος ο κλάδος να μπορεί να στηρίξει αυτά που θα βγαίνουν από την έρευνα και την καινοτομία, να μπορεί να τα εφαρμόσει. Οπότε ο, οι μελέτες αντικτύπου είναι απαραίτητες για όλες τις εταιρικές σχέσεις. Θα γίνουν σιγά σιγά. Χρειάζεται οπωσδήποτε μια αναλυτική τουλάχιστον δουλειά για κάθε μία από τις εταιρικές σχέσεις. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα εξ ονόματο τη Μαρία Γκαμπριέλ, αλλά σίγουρα η Επίτροπος θα χαρεί πολύ να είναι εδώ στην ακρόαση 18 Φεβρουαρίου. Βέβαια πρέπει να δούμε λίγο και το ε, χρονοδιάγραμμά της, την ατζέντα της, αλλά θα ήταν πολύ χαρούμενη πιστεύω να έρθει. έγιναν διάφορα σχόλια για τη συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, δεν μπορώ να σχολιάσω ακόμα, αλλά από, την, από τα σχόλια της ε, Κομισιόν και από τη, τα, ε, τα, τις δηλώσεις Προέδρου στην ΚΟΠ στη Μαδρίτη φαίνεται ότι χρειάζεται να δουλέψουμε πολύ σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας για να ε, επιτύχουμε τους ε, στόχους μας για το περιβάλλον και είναι σαφές ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κεντρικό όχημα για τη χρηματοδότηση αυτής της έρευνας. Οπότε για μένα το θέμα είναι πώς το Horizon Ευρώπη μπορεί να συνδεθεί με τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά και με το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη, το πρόγραμμα για το διάστημα, το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη, το InvestEU και με άλλους τομείς όπως η γεωργία ας πούμε, όπου η χρήση καινούριων τεχνολογιών ε, θα μπορούσε να έχει χώρο και περιθώριο. Πρέπει να επενδύσουμε στις τεχνολογίες. Έχουμε ήδη ξεκινήσει με προγράμματα σε συνεργασία με την βιομηχανία. Ε, ίσως ακολουθήσουν η αεροπορία, ο χάλιβας, άλλα επίσης. Να δούμε βασικά, βασικούς κλάδους στους οποίους θέλουμε να επιφέρουμε καινοτομία. Θα πρέπει να είναι project ισχυρού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που να έχουν όμως εξασφαλίσει και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων ε, της έρευνας. Ε, τώρα βέβαια το να κάνουμε προτάσεις για εταιρικές σχέσεις χωρίς να έχουμε προπολογισμό είναι ε, πρόβλημα. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε πριν τα θεσμικά όργανα συμφωνήσουν για το μελλοντικό προπολογισμό. Θα το δούμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις μέσα στο 2020 και είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο <clears throat> οι διαπραγματεύσεις πρέπει να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Στην αρχή του επόμενου έτους θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες επιπτώσεων, το Μάρτιο, τον Απρίλιο το πολύ, οπότε οι νομικές πράξεις ε, θα είναι έτοιμες γύρω στο καλοκαίρι. Οπότε θα Και αν ε, μέχρι τότε έχει προκύψει και συμφωνία για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Οι εταιρικέ σχέσει ε, ήδη χρηματοδοτούνται μέχρι το τέλο 2020 με πιστώσει ανάληψη υποχρεώσεων και μετά μέχρι το 2022-2024 μπορούμε να λειτουργήσουμε τον υπάρχοντα προπολογισμό αλλά η νομική δουλειά μας πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι το τέλος του 2020. Τώρα, ποιες ε, αποστολές είναι οι πιο προχωρημένες. Όπως σας είπα, είναι η αποστολή για τις πόλεις, Και νομίζω ότι από εκεί θα προκύψουν οι πρώτες συστάσεις. Το σημαντικό είναι οι αποστολές να συνδεθούν με άλλες εξελίξεις στην πολιτική μας. Θα πρέπει να προφανώς να απευθυνθούμε σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και ένα ευρύ πεδίο πολιτικών. Οι πόλεις είναι χώροι με πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλούς κατοίκους, οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη εργασίες που ήδη γίνονται και να προσθέσουμε αξία μέσω των αποστολών. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ήδη πράγματα τα οποία γίνονται στη συνεργασία της, ε, ε, της βιομηχανίας και ε, των τοπικών πληθυσμών. Οπότε πιστεύω ότι ε, για παράδειγμα, θέλω να πω ότι ε, θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη το πρόγραμμα δράση για τον καρκίνο, ε, που θα πρέπει να ενταχθεί μέσα στη δική μας δουλειά. Ο πρόεδρος μου θυμίζει ότι έχουμε κι άλλο ένα γύρο ερωτήσεων. Προσπαθώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας συνέργειες και απλοποίηση. Είναι σημαντικό θέμα, έχει ήδη γίνει πρόοδος. Να πούμε καταρχήν ότι ε, ε συζητάμε με όλα τα κράτη-μέλη, εξηγούμε πώς σκεφτόμαστε την εφαρμογή του Οριζόντας Ευρώπη, την αξιολόγηση, ε, Πώ μπορούμε να συνδέσουμε το Horizon Europe με άλλα ταμεία και παίρνουμε πολλέ απόψει. έχουμε πολύ feedback, αλλά ταυτόχρονα με αυτή τη διαδικασία βοηθάμε όλα τα κρατη να έχουν την ίδια κατανόηση των κανόνων προκειμένου να το πάρουν στα χέρια τους και να συνεχίσουν την απλοποίηση. Από το σχόλιο σας κρατώ το ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε πως η απλοποίηση μερικές φορές έχει σχέση με τη συνέχεια, δηλαδή να μην αλλάζουν οι κανόνες κάθε τόσο Προφανώς δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Θα βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε και θα διατηρήσουμε αυτά τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους. ένα ενίο σύνολο κανόνων είναι πολύ σημαντικό ε, μαζί με τους κανόνες αξιολόγησης. Αλλά και στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο συζητάμε το κατά πόσον όταν συνδυάζουμε πολλά μία και συντονίζουμε αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα, ένα ενιαίο σετ κανόνων. Θα μπορούσε αυτό να εξασφαλίσει απλοποίηση αλλά δεν είναι εύκολο. I was myself uh, also disappointed by the limited participation of civil society organizations. Και μένα με απογοήτευσε η περιορισμένη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαβούλευση. Εμείς είχαμε κάνει πολλή διαφήμιση Ταυτόχρονα όμως μην ξεχνάμε ότι η κοινωνία των πολιτών δεν συμμετείχε ποτέ στο παρελθόν, η πρώτη φορά που συμμετέχει. Πάντω η αλήθεια είναι ότι και εγώ θα ήθελα να συμμετάσχει πολύ περισσότερο η κοινωνία των πολιτών. Θα συνεχίσουμε να την ενθαρρύνουμε. Συνεργαζόμαστε με πολλές από τις οργανώσεις ομπρέλα στις Βρυξέλλες έτσι ώστε να συνσχεδιάζουμε τα προγράμματά μας με τους πολίτες. Θα θέλαμε οι πολίτες οι ίδιοι να συμμετάσχουν και όχι οι οργανώσεις τους, ε, θα το προσπαθήσουμε. Τώρα, η εφαρμογή του προγράμματος για τους κρατικούς φορείς ε, αυτό που λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά είναι το δημόσιο συμφέρον. Ο δικός μας ρόλος είναι να επιτρέψουμε στην βιομηχανία να συμμετάσχει, αλλά να τις πρόξουμε να πάει λίγο πιο πέρα. Για παράδειγμα, στην εταιρική σχέση για την πολιτική αεροπορία, η, η εταιρική αυτή σχέση ήδη δημιουργεί μεγάλα, μεγάλο όφελος με τη μείωση το, της κατανάλωσης για παράδειγμα. Ε, αλλά στο μέλλον θα χρειαστούμε όχι απλώς μεγαλύτερο προπολογισμό στην έρευνα, αλλά πραγματική καινοτομία που να είναι κάτι πραγματικά καινούριο σε σχέση με τις παλιότερες τεχνολογίες. Μόνο έτσι θα πάμε πολύ πιο μακριά. Αν μου δώσετε ένα ακόμα λεπτάκι, λέτε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα πετυχημένες στον, στο πρόγραμμα Horizon 2020. Δεν υπάρχει τίποτα στην καινούρια προσέγγιση που θα παρεμποδίζει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αντίθετο. Προσπαθούμε να διευρύνουμε τη σύνθεση των εταιρικών σχέσεων και βλέπουμε αυξημένο ενδιαφέρον πλευράς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην ε, εφαρμογή επίσης. Σε ό,τι αφορά τι αβεβαιότητε. ναι, η δημοσιονομική αβεβαιότητα υπάρχει, δεν μπορώ να προσθέσω κάτι. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, θα πρέπει να συνεργαστούμε για να μειώσουμε και τις αβεβαιότητες. Η βασική διαφορά μεταξύ του Horizon 2020 και του Horizon Ευρώπη είναι η προσπάθεια που κάνουμε να εστιάσουμε σε θέματα τα οποία είναι οριζόντια μεταξύ πολλών κλάδων. Δηλαδή, το ορίζον 2020 ήταν πολύ πιο κατακαιρματισμένο σε κλάδους, σε συγκεκριμένα κομμάτια της βιομηχανίας. Εδώ προσπαθούμε να εστιάσουμε σε θέματα που είναι πιο οριζόντια. και θα πρέπει να ξαναδούμε την, ε, το πώς συνεργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε εμείς ως Κομισιόν με τους ενδιαφερόμενους. Θα πρέπει να κατανοήσουν αυτή την καινούργια προσέγγιση και εδώ δημιουργείται καινούριο χώρος για συμπράξεις ε, και ομάδες εταιριών που θα συνεργαστούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συγκεκριμένες απαντήσεις σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Έχουμε 7 συναδέλφους που ζήτησαν τον λόγο. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε για την εκλογή σας. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες άλλες ερωτήσεις ε, για την θεσμική συνεργασία. και θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις για το νέο κομμάτι του ορίζοντα για την Ευρώπη. Από ό,τι κατάλαβα από τις ε, προηγούμενες απαντήσεις σας, πρέπει να περιμένουμε 13 ξεχωριστά νομοθετήματα που αφορούν τον προπολογισμό μέχρι το καλοκαίρι του 2020 και έχουμε μια σειρά συνεργασιών που αφορούν τα άρθρα 1 και 5 ε, που είναι στην ε, συναπόφαση και κάποια άλλα που είναι ε, δημόσιο προς ιδιωτικό τομέα που βασίζονται στο 1.7. Υπάρχουν όμως κάποιες συζητήσεις ακόμα για το αν θα είναι 1.5 ή 1.7. Θα ήθελα λοιπόν κάποιες διευκρινήσεις ειδικά όσον αφορά τις ε, ε, εταιρικές σχέσεις και αν σκοπεύετε να επεκτείνετε τον συνολικό αντίκτυπό τους ε, και συμφωνώ πλήρως βεβαίως, αλλά ποιες είναι οι συζητήσεις που κάνετε για την απόφαση αυτή, αν είναι δημόσιο με δημόσιο ή δημόσιο με ιδιωτικό τομέα και αν έχουν όλα αυτά ρυθμιστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Γκάλβες Μινιός για τους σοσιαλδημοκράτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ κύριε Πακέ που ήρθατε. Λοιπόν, έχω δύο ερωτήσεις, ε, μία για τις ε, αποστολές ε, και μία για τις εταιρικέ σχέσεις. Η πρώτη αφορά τις ε, περικοπές προπολογισμού, τις προτεραιότητες και την ε, συνέργεια. Νομίζω ότι η προσέγγιση αυτή έχει τη δυνατότητα να επιτύχει την ευθυγράμμιση των προγραμμάτων που δεν έχουν επαρκή συνέργειες. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται επαρκής ε, προϋπολογισμός, αλλιώς κινδυνεύουμε ε, να έχουμε ένα πρόγραμμα βεβαίως αλλά χωρίς, χωρίς οριζόντιες προτεραιότητες ε, που θα επιτύχουν συνέργειες. Το ερώτημά μου λοιπόν, εάν είναι αρκετά μεγάλες οι και ε, οι αποστολές θα είναι προτεραιότητα. Όλες οι αποστολές, κάποιες από αυτές. Ή θα μειώσουμε την φιλοδοξία κάποιον από αυτόν. Παραδείγματο χάρη να αναφέρατε την πιο προθυμένη εξ αυτών και ανταυτού αυτό το οποίο είχε πει η κυρία Ματσουκάτο για τις πόλεις με πολύ χαμηλές εκπομπές μπορούμε να πούμε για ηλεκτροδότηση πόλεων αυτό το οποίο προτείνουν κάποιοι κάτι το οποίο είναι πιο μετριοπαθής στόχος. Οπότε το ερώτημά μου είναι αν ε, είναι μεγάλη περικοπή του προπολογισμού, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες. Η άλλη ερώτηση αφορά μία από τις εταιρικέ ε, σχέσεις. Η αξιολόγηση αντικτύπου δεν πηγαίνει όπως ε, περιμέναμε. Παραδείγματο χάρη στην συνεργασία πρίμα και εμείς θέλουμε πράγματος χάνει να ε, μάθουμε θα είναι αντίθετη στην συνέχιση μέχρι το 2021 και να δούμε βέβαια το θέμα της ε, διαθεσιμότητας ε, του νερού και της πρόσβασης στην γεωργία στη Μεσόγειο σε μια περιοχή σημαντικά γεωπολιτική. Οπότε το ερώτημα είναι αν ισχύει αυτή η φήμη ή όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μιχαήλοβα από το Ρινιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την εκλογή σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθύντα που ήρθατε και μας παρουσιάσετε αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Εγώ θα συνεχίσω σε μια κατεύθυνση παρόμοια με αυτήν την οποία έκανε η συντονίστρια της ομάδας Ριγνιού. Αναφέρατε ήδη κάποιες από τις επιλογές με το μέσο συνδέοντας ε, την Ευρώπη με το διεθνικό πρόγραμμα και τα άλλα προγράμματα. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Ε. Στην ατζέντα εκεί των συνεργασιών και των αποστολών υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής ε, με νέα προγράμματα. Και ε, οι άλλες επιλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν να είναι αποτελεσματικός ο προπολογισμό της Ένωσης, ε, να μην υπάρχει άλλη επικάλυψη, να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα από όλα τα προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους πράσινους τρόπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας συγχαίρω και εγώ. Ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά. Έχω λοιπόν σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και κάποια σχόλια. Πώς εφαρμόζεται το πρόγραμμα ορίζοντας 2020, ε, πόσα λεφτά έχουν ήδη υπογραφεί και σε τι ποσό σκοπεύετε να φτάσετε μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Γιατί ρωτάω. Η Κομισιόν προτείνει να τεπλασιαστεί αυτό το πρόγραμμα λοιπόν. Θα πρέπει ακριβώς να βρεθούν ήδη οι πόροι για να συνεισφέρουμε σε αυτό το πρόγραμμα για να μην περικοπούν άλλα προγράμματα. πέρα έχουμε και κάποιες περιοχές συνοχής όπου χρησιμοποιούνται τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής από όχι τόσο πλούσιες χώρες και βεβαίως έχουμε αρκετά μεγάλη κατανομή για τα προγράμματα του κλίματος. Κάτι άλλο. Όταν μιλάμε για τον ορίζοντα Ευρώπη δεν θα έπρεπε να προσθεθεί κάτι ε, για το πώς θα μπορούσαμε να επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους ή να λύσουμε καλύτερα τα προβλήματα στον τομέα της ε, γεωργίας. Καθώς γνωρίζουμε ότι οι τιμές αγοράς είναι μηδενικές και έχουν πολύ, αντίκτυ... πολύ αντικό αντίκτυπο στη γεωργία. Ένα άλλο ερώτημα. το πρόγραμμα χρησιμοποιείται διαφορετικά ε, από διαφορετικές χώρες. Ε, ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν και αν ε, θα υπάρχει δυνατότητα από όλα τα καρδιμένα να χρησιμοποιήσουν επαρκώς το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ε, θα ήθελα να πω ότι το εξή. Οι επιτροποί αλλάζουν κάθε πέντε χρόνια. Και θα μπορούσε να είναι πιο σταθερή η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρίς τους γενικούς διευθυντές. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε. Και να συνεχίσετε στον ορίζοντα Ευρώπη. Λοιπόν, να σας δώσω τώρα την δυνατότητα να συνεχίσετε με αυτά τα οποία είπε ο συνέλφος Ντανίκα. Γιατί έγιναν πολλές λεπτομερείς ερωτήσεις και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το Green Deal για την Ευρώπη εξαρτάται από την επιτυχία της ε, τεχνολογίας από νέους κινητήρες, νέα τεχνολογία παραγωγής, χάλιβα, γεωργία, πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε κάποια εμπειρία λοιπόν. Εν 2000 ο κύριος Αντώνιο Γκουτιέρες, ε, πρωθυπουργός της ε, Πορτογαλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αποφάσισε την στρατηγική της Λισαβόνας για την καινοτομία. Τίποτα άλλο. Το 2010 ο πρόεδρος Φαν Ρόμπα μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε τη στρατηγική της Ευρώπης 2020. Ε, την ξεχάσαμε και αυτήν. Και δεν θα θέλαμε να χάσουμε τρίτη φορά. Έχουμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κοινοτομίας. Ε, όλα αυτά υπό την αιγίδα σας, ε, κύριε Γενική Διευθυντά. Και το τρίγωνο αυτό της γνώσης και έχουμε ακριβώ ε, την ε, καινοτομία αυτή χάρη σε ένα Ινστιτούτο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και βεβαίω διεύρυνση ε, και πολλά λεφτά για την διεύρυνση για να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη και ενδιαφέρομαι να μάθω λοιπόν ποιο είναι το όραμά σας για να χρησιμοποιηθούν τέτοιες δυνατότητες για να είμαστε νικητές το έτος 2030 πώς ε, θα το επιτύχουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Τερέζα Γκρίφιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπό την ηγεσία του Γέρζη Προσπαθήσαμε ακριβώς η Ήτρε να έχει περισσότερη προϊστάμενη αξία και ελπίζω το ίδιο να κάνουμε και τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πακέ. Πρώτα απ' όλα για τον προπολογισμό δεν έχει κανένα νόημα σε σχέση με την υγεία της ε, κοινωνίας ή των οικονομικών αντίκτυπων να κόψουμε τον προϋπολογισμό. Ερώτηση. Πώς ταιριάζει αυτό με την δίκαιη μετάβαση. Η δίκαιη μετάβαση δεν είναι απλά λεφτά. Εννοούμε μια κοινωνική προσέγγιση στην βιομηχανική πολιτική, οπότε ίσως το νόημα να μην είναι μόνο η αλλαγή δεξιοτήτων των υφιστάμενων εργαζομένων, αλλά η εκπαίδευση των νέων για να, των μικρών παιδιών σήμερα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δουλειές του μέλλοντος. Το ερώτημά μου λοιπόν αφορά την διακυβέρνηση. Μιλήσατε για το πώς θα επανασυνδεθούν οι πολίτες με την επιστήμη. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δείτε ακριβώς ε, την ε, διαχείριση της ε, Ενεργειακής Ένωσης. Το ερώτημά μου τώρα για αυτά τα οποία είπατε για την οριζόντια προσέγγιση είναι το πώς όλα αυτά θα ενσωματώσουν τη διάσταση του κλίματος ε, και του φύλου. Αλλά υπάρχει κάτι το σημαντικό το οποίο είχε ξεκινήσει στην δεκαετία του 1990. Ήμουν εγώ επικεφαλής οικονομικής ανάπτυξης για το Λίβερπουλ. Και είχαμε συνεργαστεί με τον Γκρέα Μέντος, επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης 16, για να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες του προγράμματος για το MSCI. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια καλή ιδέα, αν είχε λάμβανε τεχνική αρρωγή για να αναπτύξει αυτή την ιδέα, για να λάβει χρηματοδότηση. Οπότε το ερώτημά μου είναι, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα τώρα και να συνδεθούμε περισσότερο με τις ε, τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες. Τελευταία ερώτηση, μάλλον έχετε απάντηση, αλλά ε, μπορεί να μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο πλήρης εταίρο στο ορίζοντα. με Ευρώπη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να σας συγχαρώ την εκλογή σα και τον κύριο Πακέ, με τον οποίο μπορέσαμε να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε όταν ήταν υπεύθυνο για θέματα μεταφορών. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Πολλές ερωτήσεις υπευλήθηκαν, αλλά θα ήθελα, επανερχόμενοι στο προπολογισμό, να σας ερωτήσω αν πιστεύετε ότι η μίαση του των κονδυλίων που έχει ανακοινωθεί μπορεί να επιδεινώσει την υλοποίηση των ε, στόχων και αυτό να έχει και επιπτώσεις και στο πρόγραμμα Horizon. Δεύτερον, εάν στα πλαίσια του προγράμματος Horizon Πιστεύετε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο βάσει ποιο μηχανισμό για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αν υπάρχουν λιγότερα κονδύλια θα πρέπει να υπάρχει συνεκτικότητα, συνέπεια, αποδοτικότητα των κονδυλίων που θα έχουμε. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε ως πρότυπο να ενισχυθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε επιτυχίες όπου εφαρμόστηκε. Κατά τρίτο λόγο, θα ήθελα να σας ερωτήσω, Ποιο νομίζετε ότι μπορεί να είναι η συγκεκριμένη περίπτωση ο ρόλος των περιφερειών, διότι στα πλαίσια των στόχων που έχουμε θέσει υπάρχουν στόχοι σφαιρικοί που δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν εάν δεν συμπεριλάβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την τοπική και περιφερειακή διάσταση, αυτοδίκηση δηλαδή. Πώς νομίζετε λοιπόν ότι μπορεί να ε, το ενισχύσουμε αυτό το θέμα. Είναι κάτι το οποίο ζητούν και απαιτούν σε όλες τις δηλώσεις εξάλλου υπεύθυνη της Επιτροπής Περιφερειών. Με μεγάλη ευχαρίστηση θα ακούσω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία παρέμβαση ο κύριος Κοράου. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ε, συγχαίρω για την ε, εκλογή σας κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πακέ, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σε σχέση με την ανακοινώσεις που αφορούν το Horizon. Στο Horizon 2000 δεν μπορέσαμε να κάνουμε να συμμετάσχουν οι ΜΜΕ και οι πολίτες. Γι' αυτό το νέο πρόγραμμα τώρα Δεδομένου ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για το μέλλον της Ευρώπης και εδώ έχουμε πάρα πολλά δις, δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ένα πρόγραμμα που θα επιτρέψει στους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής της Γενικής σας Διεύθυνσης να επισκέπτονται τις διάφορες περιοχές, να συνοδεύονται από ευρωβουλευτές και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να καταστήσουν γνωστά τα προγράμματα αυτά όλα στους πολίτες. Δεύτερη ερώτηση. Το νέο πρασίνισμα, το νέο Green Deal. Κύριε Πακέ, μιλήσατε για μια πραγματική βιομηχανική επανάσταση, ώστε να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τις ε, ε, ανισότητες που υπάρχουν στη βιομηχανία. Με ποιο τρόπο θα το κάνετε αυτό, πώς θα προγραμματίσετε αυτή την μετάβαση, πώς θα την εγγυηθείτε, βάσει ποιων προγραμμάτων και σχεδίων. Τρίτον, ο ψηφιακός κόσμος και οι νέες τεχνολογίες. Όντως, πάντα υπάρχει η εμπορική πτυχή. Και εδώ διερωτόμαστε ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης σχέση με τις άλλες υπερδυνάμεις. Είπα και Κίνα. Ας μην ξεχνάμε όμως ποιες είναι οι επιπτώσεις τη ψηφιοφύσης και στην απασχόληση. Προβλέπετε κάτι, κάποια μελέτη για να Δείτε ποιος είναι ο αντίκτυπος στην, στην απασχόληση. Στην... Ε, σας ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά. Τώρα σας δίδω το λόγο 5 με 7 λεπτά και φαντάζομαι ότι έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε και στα πλαίσια του χρόνου που έχει οριστεί και να μην έχουμε καθυστήρηση. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο σύντομο από ό,τι προηγουμένω, κύριε Πρόεδρο. Όσον αφορά τι συμπράξει εταιρικέ σχέσει, κάνουμε 13 μελέτες αντικτύπων. Δεν προδικάζουν τα αποτελέσματα. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να δημιουργηθούν αυτές οι πράξεις και είδατε στην ε, στρατηγικό σχεδιασμό ότι αναφέρονται αυτά. Για καθέναν από αυτούς βλέπουμε ποιες είναι ο τρόπος εφαρμογής τους και ποιες είναι οι εναλλακτικέ λύσεις. Άρα προσπαθούμε να είμαστε αποδοτικοί, από κοινωνικοί και περιβαλλοντικής πλευράς. Ποιος είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος να καταστήσουμε αυτές τις συμπράξεις αποτελεσματικά. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα εάν θα υπάρξουν 13 προτάσεις, εάν θα καλυφθούν όλες οι, όλοι οι τομείς τους οποίους θέλουμε να καλύψουμε. Υπάρχει τα, η σύμπραξη μεταξύ ε, Ευρώπης και Αφρικής που αρχίζει από το EDCTP βάσει των άρθρων 85 και 87, στα πλαίσια του ECDP ξέρουμε ότι έχουν γίνει ήδη κάποια πράγματα και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει το κύριο σημείο της ε, σύντησης. Δεν ξέρω όμως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η ανάλυση αντικτύπου είναι, αν θέλετε, ο τρόπος με τον οποίο ξέρουμε ποιες είναι οι πολιτικές λύσεις που προτιμούμε να ακολουθήσουμε και η Επίτροπος Γκάμπριελ και άλλοι επίτροποι συνεργάζονται και θα δούμε πού ακριβώς θα καταλήξουμε. Τώρα, αν θα κάνουμε μία οριζόντια πρόταση χωριστές προπάσεις, είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε συζήτηση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει όμως μία πάρα πολύ ξεκάθαρη λύση που θα προτεθεί οριζόντια για να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις και οι λύσεις που θα ακολουθήσουμε. Δεν νομίζω ότι θα βγάλω συμπεράσματα όσον αφορά τον προπολισμό. Ακόμη δεν έχουν γίνει αποφασιστεί περικοπέ. Είστε μέλος της όλης διαδικασία ως κοινοβούλιο, άρα δεν μπορώ να πω τίποτε αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τώρα τι παραμέτρου των αποστολών. Νομίζω ότι έχουν σε κάποιο βαθμό σχέση με τον προϋπολογισμό δεδομένου ότι οι αποστολές δεν αφορούν την κοινοτομία και την έρευνα. Ο στόχος τους είναι να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα στις διάφορες κοινωνίες σε τοπικό, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πράγμα που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο από την συνεισφορά του Horizon. Βεβαίως, μεταξύ άλλων, μας επιτρέπει να έχουμε αποτελέσματα σε θέματα κοινωνίας τεχνολογιών και αν οργανωθούν σωστά και μπορέσουν να αποσπάσουν και την πολιτική προσοχή, τα κράτη-μέλη και τα ερευνητικά τους κέντρα θα θελήσουν ίσως να συμμετάσχουν. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και συμπληρωματικά κονδύλια. Θα τις ε, δείτε και θα συζητήσετε μαζί με τους υπεύθυνους του χρόνου. Οι συνέργειες, ναι. Νομίζω ότι οι συνέργειες πραγματικά αφορούν ε, ευρύτερες συζητήσεις ο, στρατηγικού χαρακτήρα και όχι μόνο για κονδύλια. Πώς ε, οργανώνεστε, πώς ε, στα πλαίσια των διαφόρων αποστολών μπορείτε να προσελκύσετε και κονδύλια από αλλού. Και βεβαίως υπάρχουν και περιορισμοί του 187 και του 185 κοινέ συμπράξεις δεν επιτρέπουν να υπέχουμε κοινού ε, κονδύλια αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και θέματα τα οποία τους επιτρέπουν να επιτρέψουν να είναι μέλος της προγραμματισμού και της προετοιμασίας το εφαρμογής των σχετικών προγραμμάτων. Και νομίζω ότι σε εκείνο το επίπεδο επίσης γίνονται και στρατηγικές συζητήσεις σε επίπεδο της Κομισιό για να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα όλων αυτών των συνεργειών. Περισσότερο από ποτέ μιλάτε αυτά τα θέματα. Επίσης, θα ήθελα να πω δύο λόγια τώρα για τα κονδύλια σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι τα διαρθρωτικά ταμεία πραγματικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και τώρα και αύριο και με αποτελεσματικό τρόπο. Αν δείτε τα αποτελέσματα, δόθηκε για το Λίβερπουλ ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Αν δω όμω τα δεδομένα, ε, της ίος ε, δημιουργούνται στην Ευρώπη περισσότερες startups, startups από ό,τι στις είπα. Είμαστε πολύ καλοί στην ε, καινοτομία, διότι τα οικοσυστήματα, στο τοπικό επίπεδο, στο και σε βιομηχανικό ε, παράγουν αποτελέσματα εξαιρετικά. Πρόκειται λοιπόν για μια προσπάθεια η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του επόμενου κύκλου. Και όσον αφορά την χορήγηση κονδυλίων σε ένα πρώτο στάδιο είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Χορηγείται και από την, και μία από τις καινοτομίες του ε, Horizon που είναι το Συμβούλιο ε, Καινοτομιών. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μια προσπάθεια ε, η οποία έχει από αυτό που γίνεται ακριβώς στο Ηνωμένο Βασίλειο και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την όλη κατάσταση με επενδύσεις κονδυλίων για τις κατάλληλες τεχνολογίες. Επίσης δίδονται και ήδη οι πόροι και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορέσαμε να δούμε και τη διάρκεια της ετήσιας διάσκεψης που γίνεται κάθε χρόνο στη Φινλανδία με 25.000 συμμετέχοντες και είδαμε ότι υπάρχει πάρα μεγάλη σχέση μεταξύ της ε, καινοτομίας, της τεχνολογίας, ε, της ε, διαχείρισης και των σταδίων μελέτης του πώς θα περάσουμε από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή κάποιων μεθόδων. Ίσως στα πλαίσια της ε, ε, συλλογής πόρων προσπαθούμε να δούμε και πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε κονδύλια απ' έξω. Ελπίζουμε όμως ότι θα μπορέσουμε έτσι να προσελκύσουμε και νέους ε, επενδυτές εκτός ε, των κονδυλίων που δίδει η Ευρώπη. Έτσι λοιπόν διασυνδέουμε τις προσπάθειες των διαθροτικών ταμείων του ε, κοινοτικού προϋπολογισμού και των κονδυλίων που προέρχονται από τις χώρες μέλη. Και τελειώνοντας θα ήθελα να αφαιρθώ και να πω κάτι για τις ε, Νομίζω ότι η κυρία Γκάμπριελ ήταν στην ακρόασή της πάρα πολύ σαφής. Θέλει να συνεχίσει να έχει ε, επίρρεια όχι μόνο στις διάφορες πρωτεύουσες αλλά και με, σε άλλες πόλεις ώστε, πόλεις ώστε να μπορέσει το πρόγραμμα αυτό να γίνει πραγματικά γνωστό σε όλους και να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Ήδη ε, για την παρουσίαση του προγραμμάτου προγράμματος προβλέπονται επισκέψεις όλες τις χώρες για να παρουσιαστεί οι κανόνες εφαρμογής και πρόκειται για εκδηλώσεις τις οποίες παρακολουθούν οι συνομιλητές μας, οι συνήθες και θέλουμε να προσελκύσουμε και περισσότερα άτομα και μπορούν έτσι και οι πολίτες να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι η ε, προσθέμενη αξία. Τώρα, η συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν κατόρθωσε να επιτύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η στρατηγική 2020 πρέπει να πω ότι ήταν ε, θετική, τώρα που ολοκληρώνεται, όσον αφορά τις επενδύσεις των κρατών σε σχέδια καινοτομίας και έρευνας, δεν έχουμε φτάσει σε στόχους. Προσπαθήσαμε να κάνουμε με τα διαρθρωτικά ταμεία και συνεχίζουμε κέντρα αριστείας, αλλά υπάρχει τώρα η αναγνώριση ότι όλα αυτά είναι σωστά και ελπίζω ότι θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια. Χρειαζόμαστε συστήματα καινοτομίας και έρευνα σε όλη την Ευρώπη, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε μία χώρα, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα για πολλές άλλες. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε συλλογικά προσπάθειες. Και η Μαρία Γκαμπριέλ κατά τη ε, διάρκεια τους θητείες της θα μπορέσει να ενημερώσει περισσότερο όλους για αυτά τα θέματα και από τις συζητήσεις σήμερα για τον Green Deal και από την Ευρωπαϊκή Πολιτική αύριο, τι συνάγουμε, ότι περισσότερο η... στον τομέα αυτό θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι το πολύ θετικό. Δεδομένου ότι πολλές κυβερνήσεις και εμείς, καθώς και εσείς και εμείς, πιστεύουμε ότι Πρόκειται για μια κεντρική προσέγγιση που θα δώσει αποτελέσματα εντυπωσιακά και θα αποτελέσει απάντηση στις ε, προκλήσεις που τίθονται στον οικονομικό, τον κοινωνικό και άλλο. Εν πάση περιπτώσει βλέπω μεγάλη κινητοποίηση και πολιτική ενέργεια. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ που μας επισκεφτήκατε για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας, να μας κάνετε αυτή την, αυτή παρουσίαση. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με την Επίτροπο, με εσά και με τους συνεργάτες σας. Θα περάσω στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης για το πρωινό μας. Παρουσίαση από την Κομισιόν της ετήσιας έκθεσης για την ασφάλεια των ε, εργασιών, υπεράκτηνων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2017. Ο κ. Στέφαν Μόζερ είναι η επικεφαλή ε, στην ε, Γενική Διεύθυνση Ενέργεια. Θα τον καλέσω εδώ. Να σα θυμίσω ότι η διαδικασία για την ασφάλεια των υπεράκτηνων εργασιών υιοθετήθηκε το 2013 αμέσω μετά ε, το επεισόδιο της Deepwater Horizon, τη BP, στον κόλπο του Μεξικό το 2010. Ε, η έκρηξη στην πλατφόρμα ε, προκάλεσε τη βήθησή της και μια μεγάλη μόλυνση. Ε, προσπαθήσαμε με αυτή την οδηγία να αποφύγουμε τέτοιου είδους επεισόδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε περίπτωση να καταστήσουμε υπεύθυνε τις εταιρείες για οποιαδήποτε βλάβη προκαλέσουν η σημερινή ετήσια, αυτή μάλλον η ετήσια έκθεση ε, δίνει στοιχεία για τον τύπο και τον αριθμό των εγκαταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενημερώνει για τα περιστατικά τα οποία ε, ανακοινώθηκαν ε, και καταγράφηκαν. είχε προβληθεί επίσης το άρθρο 40 της οδηγίας μέχρι 19 Ιουλίου 2019 η Κομισιόν να υποβάλει λαμβάνοντα υπόψη μάλλον τι προσπάθειε και τι εμπειρίε των αρμόδιων αρχών, να αξιολογήσει την εμπειρία στην εφαρμογή της οδηγίας. Θα ήθελα να μας ενημερώσει ο κ. Μόζερ για αυτό το θέμα. Δέκα λεπτά θα του δώσω το λόγο και μετά, ανάλογα με το πόσοι θα έχουν απομείνει στην αίθουσα, θα έχουμε χρόνο και για έρωτα απαντήσεις. Κύριε Μόζερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καλημέρα σε όλους και όλες. Η οδηγία για τις υπεράκτητες εργασίες ε, είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε πολύ σοβαρά έτσι ώστε να προλάβουμε σημαντικά τυχήματα, σοβαρά τυχήματα στα ύδατά μας, ε, να και για λόγους ασφαλείας των εργαζομένων αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους. Ε, προφανώς ε, επηρεάζεται πάρα πολύ και ο τομέα του τουρισμού από τέτοιου ατυχήματα. Υπάρχουν πάνω από 500 εγκαταστάσεις ε, στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωση. ένας αριθμό που μειώνεται περίπου 50% των εγκαταστάσεων ε, τέθησαν σε λειτουργία μεταξύ του 1980 και του 2000. Πολλέ από αυτές θα καταργηθούν στο μέλλον. Ορισμένες ήδη έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Αυτό είναι ένα ε, θέμα το οποίο μας απασχολεί συχνά. Η ασφάλεια, ε, τα αποτελέσματα ασφάλειας για τις πρώτες ε, δύο ετήσιες εκθέσεις ήταν σχετικά καλά. Δεν είχαμε θανάτους καθόλου. Ορισμένες πτυχές έχουν βελτιωθεί από το 2016 στο 2017. Κάποιες έχουν χειροτερεύσει. Για παράδειγμα, η ακούσιες ε, ε, επελευθερώσεις έχουν χειροτερεύσει λίγο ε, αλλά έχουμε βελτίωση στις απώλειες ελέγχου της γεώτρησης, στις βλάβες κρίσιμων για την ασφάλεια και το περιβάλλον στοιχείων και στις με σκάφη. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να υποβάλουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Η Κομισιόν έχει δώσει το σχέδιο, το, το περίγραμμα αυτών των πληροφοριών στο πλαίσιο μιας ε, κατεφαρμογή ο, εκτελεστικής μάλλον ε, συνομικά τεξουδότηση πράξης ε, όλα τα κρατημέλη έχουν δώσει πλήρη στοιχεία για τις εγκαταστάσεις με την εξαίρεση του Ενωμένου Βασιλείου το οποίο χρησιμοποίησε ένα μια νομική εξαίρεση που προβλέπεται και είναι προσωρινή περιόρισε τις πληροφορίες στις εγκαταστάσεις οι οποίες υπο, υπόκεινται σε ε, κανονιστική ρύθμιση ε, ε αυτό το, αυτή η δυνατότητα έχει καταρριχθεί από το 2018 και μετά. Ε, ε πάντως ε, ε, ακόμα και για αυτές τις οποίες μας έδωσε είναι αρκετές, είναι 139 από τις 188 συνολικά καταστάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, οπότε είναι αρκετές για να βγάλουμε συμπεράσματα. Ε, το 2017 6 εγκαταστάσεις τέτοιες ανεκτός λειτουργίας, πέντε στο Ηνωμένο Βασιλείο και μία στην Ιταλία. Αυξάνεται αυτός ο αριθμός με το χρόνο με το χρόνο. Ε, νέες εγκαταστάσεις είχαμε μία στις κατοχώρες και μία στο Ηνωμένο Βασίλειο που ετέθησαν για πρώτη φορά σε λειτουργία και υπάρχουν, υπάρχουν και μετακινήσεις μία, μία συγκεκριμένη Η τάση είναι στη συνολική παραγωγή, είναι μείωση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον Ατλαντικό και την Βόρεια ε, θάλασσα. Στη Μεσόγειο η Ιταλία είναι ο πιο σημαντικός παραγωγός, αλλά και η Κροατία και ορισμένες άλλες χώρες έχουν σκοπό να ξεκινήσουν παραγωγή, το μελετούν. Ορισμένες εξελίξεις στη Μαύρη Θάλασσα, έχουμε τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, αλλά κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο με την Κύπρο και ορισμένους από τους γειτονές μας, το Ισραήλ και την Αίγυπτο και με αυτούς έχουμε σημαντικά, έχουμε πολύ καλή συνεργασία προκειμένου ε, να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές και να εξασφαλίσουμε ότι η δική μας εμπειρία θα τουλάχιστον θα είναι διαθέσιμη για αυτές τις ε, χώρες, για αυτούς τους ε, γείτονες έτσι ώστε να τη χρησιμοποιήσουν αν θέλουν. Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα σύμφωνα με την οδηγία να επιθεωρούν τακτικά τις εγκαταστάσεις και όσο περισσότερε εγκαταστάσει έχει κανεί, τόσο περισσότερου ελέγχου θα πρέπει να πραγματοποιεί, όσο περισσότερε επιθεωρήσει. Η έκθεση δίνει πληροφορίε για τον αριθμό των επιθεωρήσεων που έγιναν. Να σα πω όμω ότι σε ό,τι αφορά τα ατυχήματα, για παράδειγμα, θα πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στα συμβάντα προ αναφορά και στα σοβαρά ατυχήματα. Τα σοβαρά ατυχήματα είναι ε, περιστατικά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρές ε, σωματικές ζημιές, ε, ακόμα και αν δεν το κάνουν. Ευτυχώς δεν είχαμε καθόλου θάνατο στο 16-17, παρόλα αυτά Είχαμε δύο σοβαρά ατυχήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα στι κατοχώρε και ένα στη Δανία. Ε, ατυχήματα τα οποία είχαν τη δυνατότητα, ενήχαν δηλαδή τον κίνδυνο να προκαλέσουν θανάτου ή ε, σοβαρού τραυματισμού. Θα πρέπει λοιπόν ιδιαίτερα αυτέ οι χώρε να ε, εξάγουν τα συμπεράσματά του, τα κατάλληλα συμπεράσματα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι αιτίε αυτών των περιστατικών. Ο αριθμό των ε, που σα αναφορά ε, είναι πιο υψηλό προφανώ, αλλά αυτά είναι λιγότερα σημαντικά. Είναι 13 συνολικά στις χώρε, 14 στη Δανία, ένα στη Βουλγαρία και ένα στην Γερμανία, καθώ επίση και 30 στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμβάντα εννοώ, ε, ε, επαναλαμβάνω προ αναφορά για το 2017. Πάντα γίνονται περιστατικά, πάντα παρουσιάζουν τέτοιου είδους περιστατικά. Το θέμα είναι ε, να μπορούμε να τα ελέγξουμε να λαμβάνουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας και να εξάγουμε συμπεράσματα και διδάγματα. Από τα συμβάντα προς αναφορά τα περισσότερα ήταν ακούσιες απελευθερώσεις. Μιλούμε για πετρέλαιο, για φυσικό αέριο που απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Συμβαίνει αυτό μερικές φορές, παρόλο που δεν είναι προφανώς επιθυμητό. Το 13% των συμβάντων που αναφορά αφορούσε απώλεια ελέγχου της γεώτρησης. Το 1,7% βλάβες κρίσιμων για την ασφάλεια και το περιβάλλον στοιχείων και 5,1% συγκρούσεις με σκάφη. Αυτά αναφέρονται από το 2017 και μετά. Το 2016 δεν τα είχαμε. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από την ποιότητα των στοιχείων που μας παρήχαν τα κράτη-μέλη. Βέβαια λυπούμεθα που εξακολουθούν να εμφανίζονται ε, αρκετά συμβάντα προς αναφορά, καθώς επίσης και μερικά λίγα ευτυχώς σοβαρά ατυχήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αν συγκρίνουμε αυτό το τομέα με τον αντίστοιχο τομέα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι η δική μας ασφάλεια δείχνει να είναι καλύτερη. Το 2017 βέβαια ποτέ δεν είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι. Θα πρέπει να βγάλουμε διδάγματα και να βελτιώσουμε τις διαδικασίες μας. Να σας πω επίσης και για την αξιολόγηση της ε, οδηγίας της ίδιας. Εξετάζουμε την επίδοση της οδηγίας συνολικά, ε, τα βασικά στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία και το πώς ε, εφαρμόζονται, το θέμα της απόσυρσης εγκαταστάσεων, ο στόχος της αξιολόγησής μας είναι να παράσχουμε ε, στοιχεία για τους εφαρμοστέους κανόνες, ποια είναι τα βασικά προβλήματα και να διαπιστώσουμε αν το συνολικό πλαίσιο είναι το επαρκές, σύμφωνα με τους στόχους μας. Το ίδιο ισχύει και για την ε, ποινική ευθύνη ή την αστική ευθύνη ε, και τις ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις ε, ολοκληρώνεται σύντομα αυτή η αξιολόγηση. Θα ετοιμάσουμε μια έκθεση την οποία θα την στείλουμε στο ε, Συμβούλιο ε, που, στο οποίο αναφερόμαστε, που είναι ένα κανονιστικό όργανο, ανεξάρτητο κανονιστικό όργανο και το δεύτερο εξάμεινο του επόμενου έτους θα είναι έτοιμο, έτοιμη η έκθεση μας δημοσίως απαντάμε σε κάποιο, με κάποιο τρόπο και στο αίτημα του Κοινοβουλίου, στις εκθέσεις μάλλον του Κοινοβουλίου της προηγούμενης θητείας για το θέμα των, της νομικής ευθύνης. και για τις αστικές και για τις ποινικές πτυχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και περιμένω τις ε, ερωτήσεις σας. Uh, uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, για τις εξηγήσεις σας ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, το ότι μειώθηκε ο αριθμός των ατυχημάτων με την εφαρμογή της οδηγίας ακριβώς για να προλάβουμε αυτές τις ατυχείς καταστάσεις και είναι σημαντικό ακριβώς ε, να δούμε και τα κράτη-μέλη. Γεγονός είναι ότι δεν πάνε όλα στην ίδια κατεύθυνση και βέβαια να παραμείνουμε σε αυτόν τον ε, διάλογο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που θα ήθελαν να παρέμβουν. Μία παρέμβαση. Ναι, παρακαλώ. ο συνάδελφος από τους Πράσινους. Ε, πρώτα απ' όλα κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια λέει ο κύριο Μπλό. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Η γενική ερώτηση είναι... Ε, θέλουμε βεβαίω να παραμείνουμε ευθυγραμμισμένοι με τη Συμφωνία των Παρισίων και τον στόχο που έχουμε και η Κομισιόν λέει ότι θέλει και είναι ένα γενικό θέμα για την Κομισιόν υπάρχει σε κάθε μία από τις επιστολές της κυρίας Φόντερ Λάιν πως ε, ε, Βεβαίω, δικαιολογείται το ότι θα υπάρχουν σε εξορίξεις αερίου και πετρελαίου από τα κράτη-μέλη. Και το άλλο το προβληματικό θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να βελτιωθούν στην οδηγία. Μιλήσατε για την ευθύνη. Η οδηγία λοιπόν δεν προβλέπει οι εταιρείε να έχουν ε, τις ε, πλήρεις δυνατότητες να πληρώσουν το κόστος. Ε, μετά μιλήσατε για τις εκπομπές ε, μεθανίου που γνωρίζουμε ότι το μεθάνιο είναι 80 φορές πιο επικίνδυνο για το κλίμα από το διοξείδιο του άνθρακα και βεβαίως η αξιολόγηση γίνεται τον Ιούλιο και θα θέλαμε να μάθουμε γιατί δεν καταφέρατε να επιτύχετε την ε, προθεσμία και να υπάρξει μια αναθεώρηση της οδηγίας για να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία δεν έχουμε ακόμα δει. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω πόσο θα χρειαστεί να περιμένει ακόμα το Κοινοβούλιο για την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της ε, οδηγίας που πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστώ κύριε Μπλός, ε, κύρια Ένστα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η οδηγία, σε αυτό νομίζω συμφωνούμε. Την ε, σημαντικό θέμα. Είπατε ήδη το τι πρέπει να γίνει και το τι έχει αλλάξει. Μας είπατε ότι όλα είναι καλά. Λοιπόν, κάνατε μια αξιολόγηση και μας είπατε ότι κάποια πράγματα πρέπει να διορθωθούν. Παραδείγματος χάρη το ότι τα περιστατικά θεωρούνται σιβαρά μόνο αν υπάρχουν νεκροί τραυματίες. Υπάρχουν όμως ε, περιστατικά ρήπανσης ε, του περιβάλλοντος των ακτών χωρίς να υπάρχει τραυματισμός ή θάνατος. Πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό το θέμα. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη εφαρμογή, κάτι το οποίο δεν γίνεται με την υφιστάμενη οδηγία. Είπατε κάποια πράγματα. Για μένα λοιπόν είναι ακόμα ανοιχτό το ερώτημα του πώς θα αντιμετωπίσετε τη ρήπανση του περιβάλλοντος, πώς θα πρέπει να ρυθμίσετε καλύτερα στην οδηγία, τι μπορείτε να μας πείτε σχετικά Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες ε, ερωτήσεις. Να ζητήσω λοιπόν τον κύριο Μόζερ να απαντήσει στις ε, συγκεκριμένες αυτές ερωτήσεις και παρεμβάσεις και βεβαίω ε, αν χρειάζεται να βγάλει και τα τελικά συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, προς τον κύριο Μπλώση για τη Συμφωνία των Παρισίων. Η Κομισιόν ε, βεβαίως είναι προσιλωμένη στην ε, απομακρυνσία από τον άνθρακα, την εφαρμογή της, του πράσινου deal, την αναβάθμιση του επίπεδου φιλοδοξίας και βεβαίως αντιμετωπίζουμε εδώ πέρα την υφιστάμενη δομή του τομέα της ενέργειας που οπωσδήποτε δεν θα είναι έτσι στο μέλλον όσο το πετρέλαιο και το αέριο παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φροντίσουμε το θέμα της ασφάλειας. Οπότε αυτή είναι μια πτυχή που πρέπει να ακολουθήσουμε πολύ σοβαρά. Η άλλη πτυχή είναι το πώς ε, θα φροντίσουμε το σύστημα αυτό ε, να ανταποκρίνεται στους ε, στόχους που θέτουμε εμείς σύμφωνα με την Συμφωνία των Παρισίων και να συνεργαστούμε και με τους διεθνείς εταίρους μας. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα να είμαστε φιλόδοξοι, δηλαδή να πάμε προς μια οικονομία ουδέτερη ως προς το κλίμα, αλλά να συνεργαστούμε και με τους διεθνείς εταίρους και να φροντίσουμε εσωτερικά εντός της Ένωσης να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει για την υφιστάμενη παραγωγή που επίσης λαμβάνει η χώρα και σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Πρέπει λοιπόν να δούμε το τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Κάνουμε την αξιολόγηση αυτή τη στιγμή, αξιολόγηση η οποία φροντίζει να συνδυάσει τα διάφορα επιχειρήματα και δεν έχει ακόμα δεσμεύσει την Κομισιόν ως θεσμικό όργανο να κάνει κάποια πράγματα και από αυτής της βάσης μπορεί η Κομισιόν να αποφασίσει Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση άρα της, νομοθεσίας του μέλλον. Αναφέρατε την προθεσμία τον Ιούλιο που μας πέρασε και πράγματι λυπούμαστε για το ότι δεν ε, την προλάβαμε και ζητώ συγγνώμη λόγος ήταν τα δεδομένα. Δεν είχαμε επαρκή δεδομένα, είπαμε ότι πρώτα πρέπει να προέχει η ποιότητα και προτιμήσαμε να περάσει λίγο παραπάνω χρόνος για να έχουμε τα κατάλληλα στοιχεία και δεδομένα και πρέπει να πούμε επίσης ότι υπήρχε μια αλλαγή της ε, Κομισιόν οπότε δεν ήταν ίσως η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και άρα θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε το να περιμένουμε λίγο για να έχουμε μια αξιολόγηση υψηλότερης ε, ποιότητας. Βεβαίω είχαμε και διαβουλεύσεις ε, με όλου τους ενδιαφερόμενους, με όλα τα κράτη-μέλη. Ε, Βεβαίω ε, δεν τα λαμβάνουμε όλα με την πρώτη, έπρεπε να τα ζητήσουμε. Ε, τώρα για την κυρία Έρνστ. Πραγματικά κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα ακόμα στην αξιολόγηση το θέμα της ε, αστικής ευθύνης εκεί πέρα πρέπει να αξιολογήσουμε πράγματι το τι υπάρχει, ποιο είναι το πλεονέκτημα του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν μπορούμε να μείνουμε στα εθνικά συστήματα αστικής ευθύνης. Ε, Αντιλαμβάνουμε αυτό το οποίο λέτε για τα σοβαρά ατυχήματα και το τι είναι σοβαρό ατύχημα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ε, νεκρούς ή τραυματίες. Βεβαίως μπορούμε να το ορίσουμε ευρύτερα, αντιλαμβάνουμε αυτό το οποίο λέτε. Ή μπορεί η ρήπανση να θεωρηθεί σοβαρό ατύχημα, είναι θέμα ορισμού. Και οπωσδήποτε θα έστελνε και ένα χρήσιμο μήνυμα, το παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Η πρακτική συνέπεια όμως ε, δεν διαφέρει πολύ γιατί και τα κράτη-μέλη παίρνουν σοβαρά και πρέπει να αντιμετωπίσουν όλα τα συμβάντα τα οποία αναφέρονται. Οπότε οτιδήποτε αναφέρεται πρέπει να πάει σε μια αξιολόγηση και πρέπει να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη με τη βιομηχανία για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. ή Ο κίνδυνος ε, τουλάχιστον Και βεβαίω ο κίνδυνο ε, για τέτοια συμβάντα μειώνεται με τον χρόνο. Όπω είπα, συνεργαζόμαστε με του ειδικού των κρατών μελών, οι αρχέ, ε, επί της αρχής είναι ανοιχτέ να συζητήσουμε τέτοια πράγματα. Ειδικά όσον αφορά την ασφάλεια υπεράκτιων εγκαταστάσεων. Συνολικά μπορούμε να πούμε πως η οδηγία είναι κατάλληλη για τον σκοπό της. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο στο μέλλον θα γίνει αξιολόγηση και θα δούμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ε, ευχαριστώ. Ε, ένα σύντομο σχόλιο γιατί έχουμε χρόνο ακόμα. Ο κύριος Μπλος ε, ζήτησε να επανέλθει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την δυνατότητα που μου δίνετε να ρωτήσω ξανά ε, εάν κατάλαβα καλά, η αναθεώρηση της ε, οδηγίας ε, θα έπρεπε να έχει γίνει τον Ιούλιο ή και πιο πριν μπορείτε τώρα να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα έχει ολοκληρωθεί γιατί το παλιό χρονοδιάγραμμα δεν τηρήθηκε οπότε υπάρχει κάποιο νέο χρονοδιάγραμμα αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση ευχαριστώ Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι η αναθεώρηση σημαίνει να δούμε το πώς λειτουργεί η οδηγία. Πρέπει λοιπόν να γίνει πρώτα απ' όλα η αξιολόγηση και θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί με τον Ιούλιο. Δεν έγινε και ζητώ συγγνώμη, εξήγησα τους λόγους. Και στη δεύτερη φάση θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση αντικτύπου. Αν αποφασιστεί ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση της οδηγίας, αυτό απαιτεί μετά συζήτηση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εντός της Κομισιόν για να δούμε αν η Κομισιόν θέλει να προτείνει μια νομοθετική πρόταση. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα μιλάμε για το δεύτερο εξάμεινο του επόμενου έτους και μετά από τη συζήτηση θα δούμε αν θα υπάρξει μια αξιολόγηση αντικτύπου. Ε, τώρα θα δούμε βεβαίως τι αντίκτυπο θα έχει ανάλογα με τις ερωτήσεις ε, ε, που θα μας έρχονται για περαιτέρω διευκρινήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε και για τις εξηγήσει. Θα θέλουμε να δούμε την επιτάχυνση της ε, διαδικασίας. Αυτά πρέπει να γίνουν σωστά. Βεβαίως ε, το μήνυμά μας ε, ε, είναι αυτό. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους, ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Λοιπόν, τα λέμε στις 2.30 ώρα.